Συνάδελφοι, καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε, γιατί προβλεπόταν η σα στις 9. Υπάρχει αμοιβαιότητα στους διαμόσου διαγωνισμούς ως θέμα, αλλά δεν θα συζητηθεί τώρα. Ο κύριος Κάσπαρη ετοιμάζει το έγγραφο εργασία του ακόμα και θα του δώσουμε ευθύ αμέσω το λόγο για να παρουσιάσει το γραπτό έγγραφο εργασία του και μετά θα προχωρήσουμε. Θα συζητήσουμε μεταξύ, μεταξύ μας με την ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Κάσπαρη, έχετε το λόγο. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ που σήμερα μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το έγγραφο εργασία. Προσπάθησα σε αυτό το κείμενο να συνεψίσω ορισμένα από τα θέματα που επανήλθαν στις συζητήσεις την περασμένες εβδομάδε και στην Επιτροπή υπάρχουν ορισμένα μέλη τα οποία θέλουν να απορρίψουν συνολικά αυτή την πρόταση της Επιτροπής και υπάρχουν και κάποια άλλα μέλη της Επιτροπής που θέλουν να ασχοληθούν με αυτή την πρόταση ως προς το περιεχόμενό της η δική μου πρόταση ήταν ε, τα άρθρα, ότι τα άρθρα 8 και 10 ε, τα οποία δεν τίθεται να αφιβόλω από κανένα μέλος να μην συμπελθούν στη συζήτηση και να συζητήσουμε τα υπόλοιπα θέματα. Τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν την περασμένη εβδομάδα ε, και νομίζω στο πλαίσιο της ακρόασης δεν δόθηκε απάντηση στην ερώτηση πόσο ανοιχτέ είναι οι αγορέ δημοσίων συμβάσεων ε, εντό Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τι αγορέ τρίτων χωρών. Δεν δόθηκε επαρκή απάντηση λοιπόν και χαίρομαι που το τμήμα αξιολόγηση αντικτύπου ε, ασχολείται με το θέμα αυτό γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή βάση επί τη οποία τελικά να ψηφίσουμε αυτή την πρόταση. Δεύτερον, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι ορισμένες χώρες μέλη έχουν ρυθμίσεις και νόμους ε, βάσει των οποίων μπορεί κανείς να εξαιρέσει κάποιους παρόχους από τις τρίτες χώρες, αλλά υπάρχει από τη, η αιτιολογική σκέψη 18 ε, της Κομισιόν που λέει ότι εάν αυτό εφαρμοστεί, στην πράξη θα ε, τεθούν εκτός ισχύω οι εθνικές ρυθμίσεις. Αλλά δυστυχώς ε, στις περαιτέρω διατάξεις του κανονισμού ε, δεν περιλαμβάνεται αυτή η πρόταση. Η δική μου πρόταση είναι προς εκείνους οι οποίοι θεωρούν ότι είναι μια προστατευτική παρέμβαση ότι όταν τεθεί σε ισχύ η ευρωπαϊκή εφαρμογή θα καταργηθούν οι εθνικές ε, διατάξεις και με τον τρόπο αυτό θα έχουμε μια ξεκάθαρη προσέγγιση του ώστε να εφαρμόσουμε την εμπορική μας πολιτική. Επίσης το θέμα κατά πόσο βοηθάει στο άνοιγμα των αγορών ή πρόκειται εδώ για ένα προστατευτικό μέτρο. Και έχω την εντύπωση ότι η εκτίμηση αντικτύπου της Κομισιόν καθώς και κρόασε εδώ στην Επιτροπή δεν ε, έδωσε μια οριστική απάντηση σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό κατά την άποψή μου όμως τόσο θα ήταν εσφαλμένο να πούμε ότι απορρίπτουμε συνολικά ε, την πρόταση της Επιτροπής. Η δική μου πρόταση θα ήταν να σκεφτούμε σε ποιο βαθμό θέλουμε να θεσπίσουμε, να συμπεριλάβουμε μια ρήτρα επανέξέταση στον κανονισμό ως ε, πρόταση Προ όλου εκείνου που είναι επιφυλακτικοί έναντι στο θέμα αυτό συνολικά, δηλαδή να του πούμε α το δοκιμάσουμε αρχικά και η Κομισιόν στην εισαγωγή ε, στο σχέδιο κανονισμού είχε πει ότι θέλει να συμπεριληφθεί μια ρήτρα επανεξέταση, η οποία όμω ε, αργότερα δεν εμφανίζεται στα επιμέρου άρθρα. Γι' αυτό θα, εγώ, η δική μου πρόταση είναι να συμπεριληφθεί μια ρήτρα επανεξέτασης. Η δική μου πρόταση είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον υποβληθεί το, η δεύτερη έκθεση, γιατί θέλει κάθε τρία χρόνια η Κομισιόν να υποβάλει μία έκθεση να τεκμηριώσει γιατί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν χρειάζεται αλλαγή του κανονισμού ή ε, ε, πρόκειται να καταθέσει μια πρόταση ε, τροποποίησης μετά από έξι χρόνια. Έτσι λοιπόν ε, θα έχουμε είτε κάποιες τροποποίησεις είτε κάποια επαρκή επιχειρήματα για το ότι δεν ε, χρειάζονται ε, αιτιολογήσεις. Και με τον τρόπο αυτό η Κομισιόν θα εκπληρώσει τα καθήκοντά της σωστά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προσέξουμε να μην ζημιώσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες στη δική τους ανάπτυξη. Γι' αυτό η πρότασή μου προς εκείνους που θέλουν εδώ να εκπροσωπήσουν ε, με έμφαση τα, κριτήρια, τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών, να συμπεριλάβουμε τα κριτήρια της ε, Παγκόσμιας ε, Τράπεζας και να σκεφτούμε ποιες αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία, του ώστε να μην υπάρξουν μειονεκτήματα για αυτές. Ε, Τέλο, 5. Πώ μπορούμε να πετύχουμε το εφέ της μόχλευσης. Εδώ ε, πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι ε, στο άρθρο 6 προβλέπεται οι αναθέτουσες αρχές να μπορούν να αποφασίσουν κατά πόσο ε, θέλουν να αποκλείσουν παρόχους τρίτων χωρών ε, στο πλαίσιο της προκήρυξης και αν παρόλα αυτά υποβάλλουν ε, αίτηση ε, αυτή η πάροχη να αποφασίσει η Κομισιόν. Αλλά με τον τρόπο αυτό δεν έχουμε μια προβλικά αυστηρή ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, αλλά είναι οι ίδιες οι πόλεις και οι περιφέρειες αυτές που μπορούν να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις και μπορούν να υπάρξουν ορισμένες ε, κοινότητες που θέλουν να αποκλείσουν ε, κάποιο πάραχο... ενώ κάποιες ε, άλλες πόλεις ή δήμοι θέλουν να τον συμπεριλάβουν. Και έτσι υπάρχει μια ευελιξία. Δεν πρόκειται για μια αυστηρή εμπορική πολιτική και δεν θα έχουμε το εφέ της ε, μόχλευσης. Γι' αυτό η πρόταση είναι να συμπεριλάβουμε το άρθρο 6, αλλά ε, μόνο εφόσον κινηθεί η διαδικασία 8 ε, και 10, τότε να μπορούν οι κοινότητες να προσφύγουν στο άρθρο 6 και να αποκλείσουν παρόχους από αυτές τις χώρες. Τέλος, ε, όσον αφορά το άρθρο 3 και την προκήρυξη διαγωνισμών, υπάρχει η πρόταση της Επιτροπής ε, να μπορούν ε, να δέχονται οι κοινότητες σε μόνο πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις παρόχους τρίτων χωρών. Αλλά η δική μου πρόταση είναι να μην υπονομευθεί συνολικά η κοινή ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική και να μην ισχύσει κάτι τέτοιο. Ε, Κατά πάσα πιθανότητα μέχρι τη συνεδρίαση του Ιωνίου θα έχουμε τα αποτελέσματα της ε, έρευνας, ε, της μελέτης αντικτύπου ε, στο Κοινοβούλιο και εντωμεταξύ υπάρχει η επίκειται και η τοποθέτηση της νομικής υπηρεσίας και δική μου πρόταση θα ήταν να αξιοποιήσουμε σήμερα την δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το κείμενο και τον ε, Ιούνιο ε, θα έχουμε και τα κείμενα από την Νομική Επιτροπή και τις μελέτες αντικτύπου και θα μπορέσουμε να ε, αναφερθούμε σε αυτά. Λοιπόν, όπως σας είπα, προσπάθησα να μέσω της ρήτρας επανεξέτασης και της ε, ε, κατάργησης των εθνικών ρυθμίσεων να άρω τις επιφυλάξεις ορισμένων. Επίσης ε, προσπάθησα να ικανοποιήσω επίσης τα ενδιαφέροντα εκείνων οι οποίοι θέλουν να περισπιστούν τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών. Και θα χαρώ εάν πραγματικά έχουμε μια πλατιά, πλειοψηφία για το θέμα αυτό, γιατί στο Συμβούλιο δεν υπάρχει αρκετή διάθεση να συζητηθεί αυτό το θέμα. Γι' αυτό θα ήθελα εμείς στο Κοινοβούλιο να μπορέσουμε να κερδίσουμε μια πλατιά πλειοψηφία για το θέμα αυτό, να μπορέσουμε στη συνέχεια να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοδομητική παρουσίαση του εγγράφου εργασία. Και τώρα να ακούσουμε του πιο συζητητέ, ο κύριο Λάγκε, από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντάνιλ. Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στο τελευταίο σημείο το οποίο ανέφερε και να το τονίσω ιδιαίτερω. Εάν συμφωνούμε για το ότι ε, θέλουμε μια τέτοια είδου νομοθεσία, θα πρέπει πράγματι να φροντίσουμε ούτω ώστε στο Κοινοβούλιο να κερδίσουμε μια ή δυνατόν πλατιά πλειοψηφία για να μπορέσουμε να περιλάβουμε τις διάφορες ε, οπτικές γωνίες, αλλιώς δεν θα κατορθώσουμε να έχουμε μια πλειοψηφία στις, ε, για να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο γιατί θα υπάρξει μια διάσπαση και εντός του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω αυτή την προσέγγιση ρητά, να προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε τις ε, διάφορες απόψεις, ούτως ώστε να υπάρξει μια πρόταση που να την χάνει ε, μεγάλης ε, πλατιάς αποδοχής για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες τέτοιες προτάσεις έναντι του Συμβουλίου, ούτω ώστε να κατορθώσουμε να μεταγράψουμε την νομοθεσία αυτή στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Και εδώ είναι ορισμένα σημεία σημαντικά, τα οποία στηρίζουμε. Για παράδειγμα, το θέμα μιας διαφοροποίησης, μιας διαφοροποιημένης τοποθέτησης έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών και εδώ πραγματικά στηρίζουμε ρητά την ε, εφαρμογή των κριτηρίων του GSP και όπου υπάρχουν πραγματικά διαφορές μεταξύ των ε, επιμέρους αναπτυσσόμενων ε, χωρών. Επίσης το θέμα της διασύνδεσης του άρθρου 6 με το άρθρο 10. Θεωρώ ότι και αυτό έχει νόημα, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε Ε, μια σωστή ε, επεξεργασία, ε, σωστή αντιμετώπιση του θέματος των εξαιρέσεων πάντοτε σε διασύνδεση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και όσον αφορά το θέμα της, των προδιαγραφών, εδώ βεβαίως πρόκειται για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, γιατί σε πολλούς ε, τομείς υπονομεύονται αυτές οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές και οδηγούν σε μια αθέμητη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Μέχρι στιγμής την ε, οδηγία για την ε, ανάθεση έργων έχουμε μια διασύνδεση με το άρθρο 59 και ίσως θα μπορούσαμε και εδώ να συμπεριλάβουμε μια αντίστοιχη διατύπωση, δηλαδή ότι κατά τον έλεγχο μέσω της Επιτροπής να συμπεριλαμβάνονται αυτά τα κριτήρια ως καθοριστικά για τον έλεγχο. Και βεβαίως ε, κατά την αξιολόγηση της ε, Επιτροπής των διαφόρων προτάσεων να συμπεριλαμβάνονται υπόψη αυτά ακριβώς τα κριτήρια το ερώτημα της ε, αναθεώρησης, ε, της επανεξέτασης μάλλον, ε, θεωρώ επίσης ότι μπορούμε να το στηρίξουμε και μπορούμε να διατυπώσουμε κάποιες βραχύτερες προθεσμίες, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε κάποιες αναπροσαρμογές αργότερα και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σωστό μήνυμα προς το Συμβούλιο, δηλαδή ότι θέλουμε να έχουμε μια αρκετά επικοδομητική στάση. Επίσης το θέμα αυτών των 5 εκατομμυρίων, κατά πόσο αυτό είναι το σωστό κατόφλι ή δεν θα πρέπει να κάνει κανείς κάποιες ε, διαφοροποίησεις ανάλογα με τις επιδόσεις. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το πανεξετάσουμε αυτό στην εξέλιξη. Αυτά είναι τα πρώτα μου σχόλια σε αυτό το πραγματικά πολύ ε, γόνιμο κείμενο εργασίας. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω άλλε και να είναι εδώ. Όμω άλλοι συνάδελφοι, αν θέλουν το λόγο, α τον ζητήσουν. Ε, θα ζητήσω συγγνώμη που δεν είναι εδώ ο Χέμεν. Απλώς ακούγοντας, Δανιέλος, ε, όσα είναι ισόρροπη η προσέγγιση. Και θέλω να μιλήσω και να εκφράσω την προσωπική μου άποψη. Νομίζω θα συμφωνήσουν οι συνάδελφοι της ομάδας μου ότι έχει εκφράσει επικοδομητική στάση εδώ και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εντατικά. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Σλέγκερμιλ που είναι μαζί μα. Ναι, εδώ είστε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την συνολικά θετική πρόσληψη και θετική στάση που έχει τηρήσει ως τώρα το Κοινοβούλιο. Ευθύς εξ αρχή είχαμε πει ότι από τη δική μας πλευρά Είμαστε ανοιχτοί στο να εξετάσουμε τις απόψει που θα ακουστούν εδώ και με αυτή τη διάθεση ήρθαμε στις διαπραγματεύσει, τη σημερινή συζήτηση. Θέλουμε να υπερβούμε κάποιες από τις φυλάξει που έχουν ακουστεί κατά τη ε, έγκρισης ενό τέτοιου μέσου και τις ανησυχίες που εκφράζονται για την ανάπτυξη σε σχέση με το όργανο αυτό. Τα αντιμετωπίζουμε με οικοδομητική στάση και αυτό που μπορώ να προσφέρω εγώ και οι συνάδελφοι από την Γενική Διεύθυνση Αγοράς είναι μια προκαταρκτική αντίδραση για κάποιες από τις προτάσεις που ακούστηκαν. Ίσως να ξεκινήσω με κάτι που ακούγεται από καιρό. Το πρώτο σημείο στο οποίο στάθηκε ο κ. Κάσπαρη. Δηλαδή το πόσο θα ανοίξουν οι αγορές και τη μελέτη αντικτύπου. Νομίζω ότι εδώ βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση. Δεν είναι τέλεια τα πράγματα και από την άποψη της στατιστικής, όπου δεν εξετάζεται πάντοτε από τους στατιστικολόγους το περιεχόμενο και έτσι χάνουμε γνώσεις νομικού χαρακτήρα. Δεν σημαίνει ότι όλες οι δημόσιες συμβάσεις λοιπόν οργανώνονται, αλλά κάποιοι χάνουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προμήθειες. Πρέπει να δούμε λοιπόν το άνοιγμα με βάση τις διεθνείς μας συμφωνίες από το ΠΟΕ και το τι περίμεναν από μας οι εταίροι μας. Δεν είναι λοιπόν αναγκαστικά το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει οι άμεσες ε, προμήθειες, οι άμεσες συμμετοχή στις προμήθειες, αλλά και δυνατότητες συμμετοχής. Μας ενδιαφέρει συνολικά το ε, υψηλό επίπεδο συμμετοχής και επίσης ε, το, ε, ο πολυεπίπεδος χαρακτήρας των περισσότερων σύγχρονων προμηθειών που θα πρέπει να μελετηθεί. Δεν είναι τόσο άμεσα τα πράγματα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτή την πολύπλοκη πραγματικότητα και γι' αυτό καταλήξαμε σε έναν απλό κανόνα. Το περιεχόμενο, ίσως να σας φαίνεται περίπλοκο κάποιες φορές, αλλά πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Να περιμένουμε λοιπόν τις μελέτες αντικτύπου για να καταλήξουμε σε περαιτέρω συμπεράσματα. Επίσης, σημειώνουμε την ιδέα ότι θα πρέπει να είμαστε σαφέστεροι για τα, τα μέτρα των κρατών μελών σε σχέση με το άρθρο 18 και 5. Η πρώτη μου αντίδραση είναι να γίνει το άρθρο 5 αρκετά εύληπτο μόνη περίπτωση όπου θα μπορούν τα κρατημέλη να λάβουν μέτρα. Νομίζω οι νομικοί εμπειρογνωμονές στηρίζουν αυτή την άποψη, αλλά καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι ακόμα δεν είναι τόσο σαφές, καθώς επιτάσσει να μην, γίνονται κάποια πράγματα, να μην γίνονται κάποια πράγματα κρατημέλη. Θα το μελετήσουμε όμως για να δούμε πώς μπορεί να διατυπωθεί καλύτερα. Έπειτα έχουμε την πρόταση για τη ρήτρα αναθεώρησης. Εδώ είμαστε ανοιχτοί Πολλέ από τι νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τέτοιε ρήτρε, οπότε νομίζω ότι μπορεί κάτι να γίνει. Δεν είμαι σίγουρο. σίγουρος. Για το αστιάκι που ακούστηκε στο τέλος, για την ε, ρήτρα σταδιακής κατάργησης. Για την ώρα δεν έχει συμπεριληφθεί στην ε, νομοθετική πρόταση. Θα πρέπει να το δουν οι υπεύθυνε για τις προτάσεις αρχές σε μια μεταγενέστερη φάση. Νομίζω περιπλοκότερο είναι το θέμα των ε, λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Το να αποκλειστούν ή να τους δοθεί ελεύθερη πρόσβαση είναι ένα μέρος μόνο της ευρύτερης αναπτυξιακής μας πολιτικής και αυτό είναι σωστό. Τώρα, δεν ξέρω εάν θα πρέπει να προσανατολίσουμε την εφαρμογή σε μέσου εισοδήματο ή ψηλότερου εισοδήματο χώρε, θα πρέπει να εξετάσουμε τι επιπτώσει που αυτό μπορεί να έχει. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να αποκλείσουμε αγορέ που βρίσκουμε ότι ήδη έχουν προβλήματα. Μπορούμε λοιπόν να πάμε πάνω από το κατόφλι μα, αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει να πάμε και στο επίπεδο του GSP. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η μόνη λύση. Θα είναι σχετικά περίπλοκη και αυτή η επιλογή. Και τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο, διότι τα θέματα κατακραματισμού και εσωτερικής αγοράς που εκφράστηκαν για το συσχετισμό μεταξύ άρθρου 16 και 8 έχουν να κάνουν με το πώ θα διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ Ρούπερτ, ευχαριστώ όλους να συστηθώ. Λέγομαι Σταρμαέρ, είμαι διευθυντή για τις δημόσιες συμβάσει στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς από την 1η Απριλίου. Να προσθέσω λίγα λόγια για αριθμούς και δημόσιες συμβάσει και να συμπληρώσω σε είπε ο Ρούπερτ μόλι τώρα. Εντό τη εσωτερική αγορά, η δίσδυση διασυνοριακού εμπειρίου στις δημόσιες συμβάσεις είναι 1,5%. Βλέπουμε ότι μεταξύ της δυνατότητα ανοίγματο και την πραγματική απελευθέρωση είναι δύσκολο να βασιστούμε μόνο σε στατιστικά στοιχεία. Το 1,5% ως ε, ε, βαθμός διείσδυσης διασυνοριακά για το άμεσο εμπόριο μας λέει κάτι αλλά όχι πολλά διότι είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός του άμεσου εμπορίου. Πολύ θετικότερος ως προς τον βαθμό δίσδυσης. Ένα δείγμα για το πόσο παραπληκτικό είναι να βασιζόμαστε μόνο σε αριθμούς για να καταρτίζουμε πολιτικές προτάσεις. Δεύτερον, σημειώνουμε την άποψή σας και την επιμονή σας να συσχετήσουμε το 8 με το 10 και όχι με το 6. Οι φίλοι και ομολογοί σας στο Συμβούλιο φαίνεται να οδεύουν στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Θα μπορούσαν να δεχτούν και το 6 και το προτιμούν από 8 προς το 10. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε όλες τις απόψεις. Είμαστε σαφώς έτοιμοι να δούμε εάν μπορούμε να βελτιώσουμε τους συσχετισμούς του 6 με το 8 και 10 από την άλλη, αλλά φοβόμαστε ότι η εφαρμογή του άρθρου 6 ανάλογα με το αν θα εφαρμοστεί όσοι έχει το άρθρο 8 ή όχι είναι κάτι που μπορεί να πηγαίνει και πολύ μακριά και εκεί μπορεί να αντιδράσουν οι ομολογίες στο Συμβούλιο. Πάντως μελετούμε, μελετούμε και προσπαθούμε να εξεύρουμε τρόπους για να βελτιώσουμε τη συνεπή διαχείριση των δύο διαφορετικών αυτών καθεστώτων. Θα πρέπει να το συζητήσουμε και άλλο μαζί σας και θα το κάνουμε ευχαρίστως. Και πραγματικά μας ε, ικανοποιεί που σας ενδιαφέρει αυτό ιδιαίτερα και πιέζεται για να προχωρήσει. Τουλάχιστον είναι σαφής η τοποθέτησή σας και την ε, η χειρά ώστε να τον καταλάβει και το Συμβούλιο. Έτσι μπορεί να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Ευχαριστούμε και καλώς ήρθατε και στο Συμβούλιο, κύριε Αλμέιδα, και ε, στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρουσία σας είναι πάντοτε μια επικοδομητική παρουσία. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Λάγκε. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή το εξή. Το ζήτημα των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων δεν το αναφέρετε. Θα μπορούσατε να αναφερθείτε στο θέμα αυτό, να επισέλθετε. Ο συνάδελφος έχει δίκιο. Η Επιτροπή δεν αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Αν μου, κύριε Γκασπάρη, επιτρέψατε μου επίσης ένα ερώτημα προς τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αγορά για το άρθρο 6 ε, καταλαβαίνω ότι στο Συμβούλιο ε, είναι υπέρ του άρθρου 6, όχι του άρθρου 8 και 10, των άρθρων 8 και 10. Το θέμα, ωστόσο, είναι εγώ το βλέπω λάθος ή τα άρθρα 8 και 10 εξασφαλίζουν μια αυστηρή κοινή ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική μόνο εφόσον μέσω του άρθρου 10 μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιους ε, παρόχους των τρίτων χωρών, μπορούμε να έχουμε μια αποτελεσματική μόχλευση. Άρα λοιπόν το άρθρο 10 είναι βασικό εργαλείο, ενώ το άρθρο 6 εάν ε, χωρίς ε, διαδικασία μπορούν οι χώρες και οι κοινότητες κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να αποκλείουν παρόχους ε, τρίτων χωρών, τότε αυτό είναι το απολύτως ε, αντίθετο. Γιατί υπάρχει πλήρης ε, κατακαιρματισμός και κάθε χώρα, κάθε πόλη κοινότητα κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί. Άρα λοιπόν δεν έχουμε αποτελεσματική μόχλευση στην περίπτωση αυτή και δεν έχουμε μια αυστηρή ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, αλλά μπορούν να αποκλειστούν κατά βούληση οι πάροχοι. Με τον τρόπο αυτό οδηγούμαστε σε μια ε, διασπορά ε, διαφόρων ε, απόψεων και υπάρχει τον αποκλεισμό τρίτων παρόχων. Εγώ θεώρησα ότι η Κομισιόν επιθυμεί να έχουμε μια αποτελεσματική μόχλευση και μια αυστηρή ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική. δεν ξέρω, γι' αυτό το ερώτημα μου είναι έχω παρανοήσει το όλο θέμα ή μπορούμε να εξέλθουμε αυτό το αδιέξοδο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Διότι έγινε αναφορά στην εφιστάμενη εθνική νομοθεσία για περιορισμούς συμμετοχής τρίτων σε δημόσιες συμβάσεις. Έχετε τίποτε να μας πείτε γι' αυτό. Ένα κατάλογο ίσως εθνικών νομοθετικών πράξεων που θα μπορούσατε να μας μοιράσετε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε το λόγο. Για να απαντήσετε σε αυτά τα τρία ερωτήματα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώς δεν είμαστε και ανάλγητοι και ακούμε και τα επιχειρήματα που εκφράσατε. Προσπαθούμε να δούμε το σύστημα από τη σωστή οπτική γωνία. Το άρθρο 6 δίνει μια αποκεντρωμένη δυνατότητα για την ώρα. Η πρόταση βασίζεται στη συνολική θεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επιμέρους ε, αιτήσει και επιθυμίες να αποκλειστούν ε, κάποια στοιχεία. Αυτό βλέπουμε ότι δεν σας αρκεί, υπάρχουν ακόμη ασυνέπειες και το καθεξής. Είμαστε πρόθυμοι να αναζητήσουμε περισσότερη συνέπεια για το σύστημα. Ίσως το να αντιστραφεί τελείω να είναι υπερβολική λύση. Όμως, η αναπερίπτωση απόκριση είναι ίσως η ευστοχότερη σε σχέση με το χρονοβόρο και περίπλοκο όργανο να γίνονται έρευνες, να υποβάλλονται αιτήσεις. Βέβαια κάποια είδους έρευνες θα πρέπει να γίνονται και βάσει το άρθρου 6. Και θα πρέπει να υπάρχει και σοβαρό λόγο για να μπορεί ένα φορέα να το κάνει αυτό. Βέβαια, το θέμα είναι και τα πολιτικά αίτια εδώ. Και η άμεση αντίδραση προς τον κύριο Κασπάρη είναι να πούμε ναι, ότι συμφωνούμε και αυτή είναι η ευρωπαϊκή τάση. Αλλά όσο απομακρυνόμαστε από τα πολιτικά επιχειρήματα και συμφέροντα, τόσο περισσότερο τίνουμε να υιοθετήσουμε αυτή τη λύση. Θα κοιτάξουμε να ενδυναμώσουμε περισσότερο και τα δύο ανάλογα με το περιθώριο που έχουμε και αυτά θα φανούν και σε έναν ενδεχόμενο τριμερή διάλογο αργότερα. Ε, για το δεύτερο ερώτημα, τα... τις εθνικές ε, νομοθεσίες και τις εθνικές νομοθετικές πράξεις. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα, όχι αναγκαστικά συμβατά με την εμπορική πολιτική μας. Η Ισπανία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Εστονία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ε, είναι χώρες για τις οποίες έχουμε σαφή στοιχεία για το τι κάνουμε. Είναι πολύ κατακαιρματισμένα ε, τα στοιχεία. Κάποιοι δεν επιτρέπουν την άσκηση ενδικών μέσων εφόσον δεν πάρει κανείς το διαγωνισμό, δεν του ανατεθεί. Υπάρχουν διαφορετικά πάντως συστήματα και πληροφορίες είναι διαθέσιμες. Βρίσκονται στην σελίδα 90 κάτι, 96 νομίζω, της μελέτης αντικτύπου. Λίγο πολύ εκεί βέβαια έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο και θα ήθελα αυτή η συζήτηση να συνεχιστεί. Να δούμε πώ βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο απόψεων. Πάντω ενστικτοδό, μπορώ να πω ότι αυτό που πρόβαλε και ο, επιχειρητή, ο, ο είναι ένα επιχείρημα που και εμά μα βρίσκει σύμφωνο, γιατί είναι πολύ σαφέ. Το πιο δύσκολο θέμα είναι η απασχόληση και τα κοινωνικά πρότυπα. Νομίζω ότι εδώ σωστά επικεντρωνόμαστε στο θέμα της αμοιβαιότητας και στο αν οι αγορές είναι ανοιχτές. Υπάρχουν όμως και άλλα μέτρα, ούτως ή άλλως, ή όργανα, ώστε να βεβαιωθούμε ότι η συνοχή, τα περιβαλλοντικά, η κοινωνική διάσκηση, διάσταση διασταση διασφαλιζονται και δεν υπάρχουν παραβιάσεις. Δεν είναι το βασικό στοιχείο έμφασης του οργάνου που σχεδιάζουμε, αλλά μετά από τόσα ακούσαμε σήμερα, ε, για πρώτη φορά μια άποψη εκφράζεται με τέτοια σαφήνεια, μια τέτοια άποψη, Οπότε θα το εξετάσουμε και πάλι για να δούμε τι μπορεί να γίνει μετά. Αναφέρθηκε το άρθρο 15, αλλά αυτό γύρει και μια σειρά από άλλα ερωτήματα, τα οποία δεν ξέρω αν είναι έτοιμα να τα ε, απαντήσουν αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη και αν έχουμε στοιχεία της τι μας μα Ε, θα το ξαναδούμε λοιπόν. Πρόεδρος, πριν ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Κάσπαρη, η κυρία Μουσκαρντίνη μόλι έφτασε και έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος της κυρίας Μακλάρκιν, των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ήθελα να εκφράσω τη στήριξή μου στον κύριο Κάσπαρη για το εξαιρετικό του έργο και ταυτόχρονα να τονίσω ότι πολλές από τις αμφιβολίες που εκφράζονται από τον εισηγητή είναι ανησυχίες που συμμερίζεται και η κυρία Μακλάρκιν και θεωρεί ότι δεν διασκεδάστηκαν ούτε από τις τοποθετήσεις σήμερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ήθελα να μεταβιβάσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη συνάδελφο ω δήλωση. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Ο κύριο Κάσπαρη να κλείσει τη συζήτηση, παρακαλώ. Äh, ναι, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Όπω σα είπα, θα χαιρόμουν αν στην ε, προσεχή συνεδρίαση έχουμε τα κείμενα τη νομική υπηρεσία και την μελέτη αντικτύπου και στη βάση αυτή θα υποβάλω το δικό μου σχέδιο έκθεσης και ε, σε σχέση με τα σημεία τα οποία συζητήσαμε την Επιτροπή ε, θα ήθελα να ήμουν, ε, θα ήμουν ευγνώμων εάν συμπεριλαμβάνεται κάποια στοιχεία όπως είπε ο συνάδελφος κ. Λάγκε σε σχέση με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Όσον αφορά δε τις ρυθμίσεις μέσω του συστήματος γενικευμένων ε, προετοιμήσεων ε, θα σας ήμουν επίσης ε, ευγνώμων εάν μας υποβάλατε κάποιες προτάσεις σχετικά. Ευχαριστώ πολύ για τη ζήτηση και θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ. Βλέπω ότι προχωρούμε σε αυτό το άκρος επίμαχο ζήτημα. Περνάμε τώρα στο σημείο 10 της μερίσιας διάταξης καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Γνωμοδοτούμε για την Επιτροπή Άγκρη και συντάκτη γνωμοδότησης είναι ο συνάδελφο Άλμπερτ Ντε. Μάλιστα σας βλέπω. Αγαπητέ συνάδελφοι, θα σας δώσω λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε αυτή την ε, γνωμοδότηση πρόκειται για μια πρόταση για μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις εμπορικές ε, ρυθμίσεις για ορισμένα γεωργικά προϊόντα και τη μεταποίησή τους. Η συγκητής είναι ο συνάδελφος κύριος Πάολο Ντεκάστρο και εδώ πρόκειται για το άρθρο 53 παράγραφος 2 και για το άρθρο 207 και τον τρόπο εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πόσο οι σχετικές ε, νομικές βάσεις στο πλαίσιο τη κοινή γεωργική πολιτική και της κοινή εμπορική πολιτική, ε, κατά πόσο υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σε σχέση με την νομοθεσία. Εν γέννη, η προσαρμογή της σχετικής νομοθεσίας αναφέρεται στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας και της κατεξουσιδότηση πράξης ε, ε, υπάρχουν ε, λίγες κατεξουσιοδότηση πράξεις. Ωστόσο, είναι δύσκολο για το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν καταξιοδότηση πράξης της ε, Επιτροπής και να υπάρξει μια συνοχή με τον ε, κοινό κανονισμό αγοράς. Ε, θα πρέπει το προβλεπόμενο διάστημα να είναι όχι 5 λεφτά χρόνια, γιατί η κοινή οργάνωση της αγοράς θα ισχύσει με το 2000. 20, ούτως ώστε να υπάρξει μια σχετική προσαρμογή. Όπως ε, γνωρίζετε, εγώ ως συντονιστής ε, του ΕΛΚ στην Επιτροπή Γεωργίας, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής, προσπάθησα να υπάρξει μια απλοποίηση και κατάργηση των ε, γραφειοκρατικών εμποδίων. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό στις συνδαστικές ε, προτάσεις της Επιτροπής Γεωργίας να αλευθούν υπόψη. Γι' αυτό ε, την τροπολογία σε σχέση με την μείωση της γραφειοκρατίας καθώς και την απλοποίηση και τη μεγαλύτερη συνοχή στην πολιτική. Ε, η κοινή οργάνωση αγοράς δεν θα ισχύσει από το 2014 αλλά από το 2015. Εγώ ασχολήθηκα με, το, με τη μεταβατική περίοδο και υπήρξα εισηγητής εδώ και θεωρώ ότι είναι, ότι είναι σημαντικό, είναι χρήσιμο να επαναπροσαρμόσουμε αυτή την προθεσμία προθα... Ε, προσαρμογής ούτως ώστε να αποφύγουμε κάποιες αρνητικές ε, παρεμβάσεις της Επιτροπής και να μην υπάρξει μία απορρίθμιση σε σχέση με τους ε, κανόνες του εμπορίου και την κοινή οργάνωση της αγοράς. Ε, δεν θα ήθελα ωστόσο να σπαθήσω το χρόνο για αυτές τις ε, τεχνικές πτυχές. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει οι γεωργοί μας να ανταπεξέλθουν στο διεθνή ανταγωνισμό. Και εδώ υπάρχει μια σχετική απόφαση του Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο του 2010, όπου με μεγάλη πλειοψηφία τότε αποφασίσαμε όλες οι πολιτικές ομάδες ότι για την γεωργία Θέλουμε μια ποιοτική προστασία, όχι μέσω των δασμών, αλλά μέσω της θέσπισης μιας υψηλής ποιότητας. Θέλουμε προδιαγραφές για το περιβάλλον, για την προστασία των καταναλωτών, επίσης ε, κοινωνικές ε, προδιαγραφές. Και εάν ε, η Επιτροπή θέλει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω εμείς στην Επιτροπή Γεωργίας δεν θεωρούμε ότι είναι προβληματικό το ζήτημα του ανοίγματο των αγορών. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, καταρχάς από την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών, ο Μπερτ Λάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν ε, δύο άξονες της συζήτηση που δεν σχετίζονται άμεσα με την Επιτροπή Γεωργίας. Καταρχήν ε, το θέμα της διαφάνειας ότι με την ε, συνθήκη δηλαδή της Λισαβόνας έναντι του Συμβουλίου έχουμε μια διαφορετική ισορροπία δυνάμεων. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την πτυχή της διαφάνειας και καθώς και την εντονότερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων και σε ποιο βαθμό εμείς θέλουμε να τις επιτρέψουμε και σε ποιο βαθμό θέλουμε το θέλουμε να υπόκεινται στον, ε, περισσότερο στον έλεγχο του Κοινοβουλίου και τι είδους προθεσμίες θέλουμε να επιτρέψουμε, ιδιαίτερα όσον αφορά τη ροπολογία υπαριθμών 4. Και θα πρέπει εδώ να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βρούμε ένα κοινό δρόμο. Αλλά εδώ η προσέγγιση και για το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων είναι να έχουμε σαφήνεια και με έναν σεβασμό των δικαιωμάτων συμμετοχής του Κοινοβουλίου. Thank you. other request for the floor. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιο το λόγο. Αν όχι, να δώσω το λόγο σαν πρόσωπο της Κομισιόν. Θέλετε να θέσετε ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Λοιπόν, ας ακούσουμε τον κύριο Σαλβατόρε Ντακούντσο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, είναι μια τεχνική σφίσεως πρόταση όπως υπογράμμισε και η συγητή σας. Ουσιαστικά πρόκειται για την ευθυγράμμιση των εμπορικών ρυθμίσεων που αφορούν ε, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα δυνάμει των νέων κανόνων της συνθήκη της Λισαβόνας κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Δεν θέλουμε δηλαδή ως Κομισιόν να εισαγάγουμε νέα στοιχεία, αλλά να παγιώσουμε κάπως το νομικό πλαίσιο. Φυσικά τι τροπολογίες του εισηγητή θα τις λάβουμε υπόψη, ιδίω σε ό,τι αφορά την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την κατάρτιση των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Επίσης, στόχος μας είναι να έχουμε και ένα πιο αποδοτικό, αποτελεσματικό σύστημα σε ό,τι αφορά την απλούστευση των διαδικασιών. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον εισηγητή για την πολύτιμη συμβολή του. Φυσικά και είναι σημαντικό στο θέμα αυτό να έχουμε παραλληλισμό και πλήρη συνέπεια με τη μελλοντική έκβαση των διαπραγματεύσεων για την κοινή γεωργική πολιτική. Αυτό είναι σημαντικό σημείο και ήθελα να το υπογραμμίσω. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, για να κλείσει τη συζήτηση, το λόγο έχει ο εισηγητής Άλμπερντ Ντέσ. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τα θέματα του συναδέλφου Μπεντ Λάγκεν, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ πλήρως μαζί σου. Θα πρέπει να προσέξουμε ούτως ώστε κυρίως να εξασφαλθεί διαφάνεια έναντι του Κοινοβουλίου και θα πρέπει όσον αφορά τις κατεξιδότηση πράξεις να έχουμε πάντοτε τη δυνατότητα να παρέμβουμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τα πάντα όσον αφορά τη νομική βάση. Ε, είναι ένα θέμα επίσης και του προσωπικού του Κοινοβουλίου. Και ε, εδώ έχω πει στη δική μου πολιτική ομάδα θα πρέπει να κάνουμε εδώ μια γενικότερη συζήτηση. Γιατί έχω την άποψη ότι θα πρέπει να μειωθεί 5% προσωπικό από την Επιτροπή και να δοθεί στο Κοινοβούλιο για να, έχουμε, ε, να είμαστε σε ίση θέση. Γιατί με τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε την επιστολή, αποστολή που μας ανατίθεται μέσω της συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, αντιθέτως εκχωρούνται όλες οι αρμοδιότητες στην ε, Επιτροπή με τον τρόπο αυτό. Ε, θα πρέπει να έχουμε επαρκές προσωπικό για να μπορέσουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια γενική συζήτηση επί τούτου. Κατά τα άλλα, συμφωνούμε νομίζω όλες οι πολιτικές ομάδες για αυτές τις προτάσεις. Σας ευχαριστώ. Αύριο λίγη προθεσμία κατάσταση τροπολογιών διότι πιέζει ο χρόνος. Διότι δεν είμαστε εμείς η καθήλυνα νομοδιαπιτροπή, είναι η Επιτροπή Άγκρη, πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Σας ευχαριστώ και τώρα περνάμε στις ψηφοφορίες. Βέβαια προβλεπόταν ε, να ξεκινήσουν στις 10 ακριβώ. οπότε προτείνω να διακόψουμε για λίγα λεπτά και επαναρχόμεθα ακριβώς στις 10 για να μοιραστούν οι λίστες ψηφοφορίας και να ετοιμαστούν οι συνάδελφοι για την ψηφοφορία.

Είμαστε έτοιμοι. Ας ε, συνεχίσουμε την συνεδρίαση με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρώτο σημείο το οποίο θα ψηφίσουμε, πρώτη έκθεση σχέδιο έκθεση για την πρώτη ετήσια έκθεση τη Επιτροπή προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τι δραστηριότητε των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων των κρατών μελών. Έκθεση του κυρίου Ζαντό. Ξεκινούμε με τη συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 14 υπέρ. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είμαι βεβαίως. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έλεγχος. 15. 14 συγγνώμη. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Κύριε Κάσπαρη ψηφίζετε. Αποχές απορρίπτεται. Ας... Ελέγχουμε την 16, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Προπολογία 17. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είμαι βέβαιος να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για τροπολογία 18. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται τροπολογία 19. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, ελέγχουμε, εντάξει. Ελέγχουμε την 20, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επόμενη 29. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ, 36 υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε την 36 παρακαλώ, άρχισε η ψηφοφορία. 36. Πέρασε. Απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 39 η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 40, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 45, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στις συστολικές αναφορές citation, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την τροπολογία 1. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις, τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές απορριπτέται 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 8 Θέλετε να ελέγξουμε την 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία, 28 ψήφους υπέρ και μόνο μία κατά εγκρίνεται η έκθεση και συγχαίρουμε τον εισηγητή, τον Γιάννη Ζαντό. Επόμενη ψηφοφορία ε, είναι το σημείο 12. Ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας Κεντρικής Αφρικής Διαδικασία έγκρισης Υπάρχει, μάλλον υπάρχουν δύο ταυτόσιμες τροπολογίες ψηφίζουμε από κοινού. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται τελική ψηφοφορία. Στο τεφά τη σύσταση για χορήγηση έγκριση σύμφωνης γνώμη. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 24 ψήφι υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές. Επόμενη Επίσης, η στάση για τη διαδικασία συμφωνής γνώμης, παράλληλη συμφωνία, Οικονομική Επιτροπή των Εθνών. Νομίζω είναι κάποια πρώτα για τα αυτοκίνητα οχήματα. Αν δεν απατώμε, τέλος πάντων, να ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. ψηφοφορία. εγκρίνεται με 28 ψήφους υπέρ και μία αποχή. Πάντα έγκριση σύσταση για το σημείο 14 ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Ομόφωνα δεκτή με 28 ψήφους υπέρ. Σχέδιο ψηφίσματο τώρα για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με πολυμερή σύμφωνη για τις υπηρεσίες στο σημείο 15. Δικό μας ψήφισμα, είμαι ο εισηγητής από την ιδιότητά μας Προέδρου και ψηφίζουμε. Τροπολογία 11. Ψήφι υπέρ. Το ΕΛΚΑ τι κάνει. Τροπολογία 11. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14, υπέρ. Α, με συγχωρείτε. Είναι τμηματική ψήφα. Πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της 14, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε. Άρχεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα τι ψηφίζουμε. Τη 15. Μάλιστα. Τροπολογία 15. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22. Προφορική τροπολογία πράγματι από την κου εδώ. Μπορείτε να μας πείτε περί τίνος πρόκειται. Μέρφυ Θέλουμε το deplores να μετατραπεί σε regrets στα αγγλικά. Με ορισμένες πολιτικές ομάδες ε, συμφωνήσαμε να είναι λίγο πιο ήπια η διατύπωση το diplore είναι πιο έντονη ως διατύπωση. Υπήρχε ε, χθες το βράδυ αυτή η συνάντηση και η συμφωνία με το Χέλμουτ δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε και να τον ενημερώσουμε, γι' αυτό και έγινε αυτή η πρώτη. Υπάρχει πρόβλημα να κατατεθεί αυτή η προφορική τροπολογία, λέει ο πρόεδρος. Όχι, άρα ψηφίζουμε τροπολογία 22 με την προφορική τροπολογία ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 24 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 26 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 27 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε την 36. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε τη συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 37 και 38 ταυτόσιμες τροπολογίε καταπίπτουν. Καταπίπτουν. άρα που πηγαίνουν στη συμπαστική 2. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, ψήφι περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε και το τρίτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 48 κατά πιπτροπολογία, συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ. Λοιπόν, να σηκώνετε τα χέρια σας. Συμβιβαστική 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την συμβαστική 3 την ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Με δύο ομάδες δεν ε, μπορείτε να κερδίσει ψηφοφορία μόνο. Λοιπόν, η 50 έχει αποσυρθεί, άρα πηγαίνουμε... Η Σκά Κέλλερ συμφωνεί μάλιστα, άρα από 51 πάμε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το αρχικό Ψηφίζουμε χωριστά το πρωτότυπο της παραγράφου 9, δάφιο 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ...54 και 55 ψήφι υπέρ. 54 και 55 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 57 δεν ήταν αυτή, μάλιστα. Ωραία. 58 τώρα. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 65 περ κατά αποχές απορρίπτεται ελέγχουμε ελέγχουμε τον 65 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 66-67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική υπάρχουν 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τοπολογία 75. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Στα ρισάιτας τώρα, ε, σε τουλικές αναφορές. 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασης της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ποια ήταν αυτή? Η 4. Λοιπόν, επόμενη. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 8. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ελέγχουμε την 9 άρχεται η ψηφοφορία ελέγχουμε την υπαρθμόν 9 τροπολογία πέρας ψηφοφορίας κάτι πήγε καλά εδώ εγκρίνεται με πολύ μεγάλη ψηφοφορία στην 9 ε, πάμε στην 10 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στο 1, στις citations εγκρίνεται, 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε την τροπολογία 2, στην αιτιολογική αναφορά 4, citation 4. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είμαι βέβαιος να ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Τέσσερις ψήφοι υπέρ και πέντε κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Επόμενο θέμα 16, ε, συγγνώμη, εντολή για τον τριμερή διάλογο. Ο εισηγητής μας είναι ο Πέτερ Στάσνη. Ε, τροπολογία υπαριθμών 1. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την τροπολογία επαλήθευση. Άρχεται ψηφοφορία για την 11. Πέρα της ψηφοφορίας. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία επαθμών 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είμαι σίγουρος. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 4. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 25 περ, 2 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Στράσνη. Επόμενο, το επόμενο θέμα αφορά τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών ε, υποθέσεων για μια συμφωνία σύμπραξης και συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαλαισίας. Συντάκτη είναι ο Νικολό Ρινάλδη. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2. D υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία μόνο 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ και 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 και 28 έχουν αποσυρθεί 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε 25 ψήφοι υπέρ 4 κατά Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι το πέρας, η λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Και τώρα θα περάσουμε στο θέμα 18. Παρακαλώ. Καθίστε. Το θέμα 18 είναι μια γνωμοδότηση της ε, ΙΜΚΟ που είναι η αρμόδια επί της επιτροπή. Η δική μας συντάκτρια γνωμοδότησης είναι η Κριστιάνα Μουσκαρντίνη, αριστερά μου, και στην οποία δίνω το λόγο. Παρακαλώ. E Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, την προσοχή σας παρακαλώ. Προτεραιότητα στον ακούγεται έχει η ομιλήτρια. Πρόεδρε, και πάλι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που η Επιτροπή μας έχει εξετάσει επανειλημμένως με την ευκαιρία του προηγούμενου κανονισμού που όπως ξέρετε όμως πάγωσε σε επίπεδο Συμβουλίου. Σήμερα πρέπει να ασχοληθούμε με το ίδιο θέμα, αλλά το οποίο έχει λάβει ευρύτερε διαστάσει. Διότι ρητό γίνεται πια λόγο για την ασφάλεια των ε, καταναλωτών. Η ελεύθερη διακίνηση των καταναλωτικών προϊόντων, που να είναι νόμιμα και μη παραποιημένα, είναι ένα από του πυλώνε από τα θεμέλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και για να υπάρχει εμπιστοσύνη στους καταναλωτές, αλλά και για να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους να επιλέγουν και να αγοράζουν αυτά που γνωρίζουν και επιθυμούν. Η δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για τα μη εδόδημα καταναλωτικά ε, προϊόντα είναι κάτι που μέχρι τώρα ελέγχεται από τις εθνικές αρχές που υποβάλλουν τα προϊόντα σε διαφορετικούς ελέγχους με διαφορετική ερμηνεία κατά την εφαρμογή των ε, σχιουσών διατάξεων. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες αποκλήσεις ακόμη και αυτό δεν επιτρέπει την επαρκή εποπτεία και την ενοποίηση της εσωτερική αγορά. Το ίδιο και για το κόστο που επιβάλλεται στι επιχειρήσει. Ο κανονισμό είναι σίγουρα φιλόδοξο και προβλέπει διάφορε υποχρεώσει για καταναλωτέ, παραγωγού και εισαγωγή, καθώ και διανομή, με την καταγραφή των απαραίτητων πληροφοριών που θα πρέπει πάντοτε να είναι ερωτές προ του καταναλωτέ. Γι' αυτό ε, στόχος είναι η χνηλασιμότητα των προϊόντων με την ένδειξη προέλευση με βασικέ προποθέσει ώστε να διευκολύνεται η αρμοδιότητα ποιότητα των εποπτικών αρχών να μπορεί να εντοπίζεται ο τόπος παραγωγής, η καταγραφή της χώρας προέλευσης και στα πλαίσια της διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας. Όπως γνωρίζετε, ένα από τα βασικά μας προβλήματα είναι η ποιότητα των προϊόντων, η προστασία των καταναλωτών, η καταπολέμηση της παραποίησης, επειδή αντιφάσκει με τις ανάγκες της εργασιακής αγοράς, προκαλεί ανεργία και στρεβλώσεις και από οικονομικής σκοπιάς. Αυτό λοιπόν που δεν θεωρούμε με την συζήτηση που έγινε και για το όλο θέμα, αυτό που δεν θεωρούμε και ζητώ από όλους τους συνοδέλφους να μου στείλουν τις παρατηρήσεις τους, ε, αυτό που δεν θεωρούμε σημαντικό, που δεν θέλουμε μάλλον να γίνει, είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει σύγχυση στο κείμενο σε ό,τι αφορά τι κυρώσει, τα πρόστιμα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε στα πλαίσια ενό ρυθμιστικού ε, συστήματο που θα ισχύει για όλες τις χώρες και θα τις υποχρεώνει να καταδεικνύουν την ε, προέλευση, δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα αρμονισμένο σύστημα σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Ιδάλλως, οι εισαγωγείς ή οι μεταπολιτές θα πηγαίνουν να δραστηριοποιηθούν στην ευρωπαϊκή χώρα που έχει τι λιγότερε κυρώσει σε σχέση με τι υπόλοιπε. Η εναρμόνιση λοιπόν των κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σημαντική και θα πρέπει να οργανωθεί στη βάση της αξίας του εμπορεύματος, του προϊόντος, του αγαθού και την ποσότητα, των όγκο παραγωγή. Δεν ζητούμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντό εισαγωγικών να ορίσει ευρώ αναπρόστιμο, τιμή, αλλά τα κριτήρια που θα ισχύουν και θα διέπουν τι κυρώσεις και θα πρέπει να ισχύουν ομοιόμορφα σε όλες τις χώρε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. α προχωρήσουμε στα υπόλοιπα μέλη που έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Δεν βλέπω κανείς να ζητά το λόγο. Όχι, κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε τη συμπερίληψη της υποχρεωτικής ε, ένδειξη ε, προέλευση για να διασφαλιστεί η χνηλευσιμότητα των προϊόντων. Επιθυμούμε όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είχε κάνει ένα στενότερο σχετισμό στο κείμενο μεταξύ των διατάξεων για την γεωγραφική προέλευση και το σύστημα χνηλευσιμότητας. Το σύστημα εχνελασιμότητα που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή είναι αρκετά δύναμο και θεωρούμε αρκετά περιορισμένο στην εφαρμογή του, εφόσον ε, μπορεί να ισχύει μόνο για υψηλοκινδύνου προϊόντα και να εφαρμοστεί εκεί. Θέλουμε λοιπόν η Επιτροπή να καταρτήσει έναν τελεχή κατάλογο τέτοιων προϊόντων με κατεξουσιοδότε πράξει. Όμω δεν έχει παραμέτρου να... και κριτήρια για να εντοπιστούν τα προϊόντα στο ε, σώμα του κειμένου και αυτό πρέπει να γίνει ε, για να εγκριθεί από του νομοθέτε. Επίση, ο κανονισμό πρέπει να σαφεί το γεγονό ότι η εχνηλασιμότητα και το σύστημά τη θα πρέπει να εφαρμόζονται και στα εισαγόμενα προϊόντα. Οι οικονομικοί φορεί είναι υπεύθυνοι για την αποτίμηση τη συμβατότητα των προϊόντων με τι ε, απαιτήσει ασφάλεια και θα πρέπει να συμμορφώνονται με διάφορε διαδικαστικέ απαιτήσει. Πρώτα απ' όλα την εποπτεία τη αγορά. Εκεί οι αρχέ θα πρέπει να έχουν ε, ε, συστηματικότερη συμμετοχή, ώστε να είναι βέβαιε ότι οι οικονομικοί φορεί σέβονται αυτέ τι υποχρεώσει. Επιπλέον, ο κανονισμό δεν προβλέπει αναλογικά μέτρα για τον ενδεχόμενο κίνδυνο ενό προϊόντο, Θα πρέπει να δώσει ένα σαφή ορισμό για αυτό το θέμα. Ιδάλλως η αναλογικότητα των διαδικασιών ω προ τον κίνδυνο είναι τελείω ε, στη διακριτική ευχέρεια των οικονομικών φορέων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Χρειάζεται να γίνουν αλλαγέ. προκειμένου να είναι σαφέστερο, κατανοητότερο και το σύστημα εχνελασιμότητας να είναι ισχυρότερο. Any request Υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει να πάρει το λόγο εκ μέρους Επιτροπής. Ε, από τα μέλη της Επιτροπής, συγγνώμη. Ας ακούσουμε τώρα την Επιτροπή. Ποιος θα μιλήσει εκ μέρους της Επιτροπής, η κυρία Δέσποινα Σπανού ή ο κύριος Νικολόφ. Έχει, ε, Δέσποινα Σπανού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, υποθέσεις των καταναλωτών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, δίνουμε μεγάλη σημασία στο εμπόριο και στη διεθνή πτυχή διάσταση αυτής της πρότασης, έχοντας ε, κατά νου ότι πολλά προϊόντα εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίσης επειδή η διεθνής πτυχή βεβαίως έχει κρίσιμη σημασία. Όταν ε, πρόκειται για την σήμανση της προέλευσης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της εργασίας της κυρίας Μουσκαρντίνη, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η Επιτροπή δεν προτείνει κάτι το επαναστατικό, είναι κάτι το οποίο ήδη προβλέπεται από πολλές νομολογίες και έχει υπάρξει το αντικείμενο συζήτησης επί πολλά χρόνια. Βεβαίως είναι σημαντικό στοιχείο της πρότασης γιατί συνδέεται με το ζήτημα της αχνηλασιμότητας. Ε, και ε, το θέμα αυτό είναι σημαντικό στην μαθηματική διαδικασία και θεωρούμε ότι επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεων υπό το πρίσμα αυτό, γιατί ο δικός μας στόχος όταν προτείναμε αυτό το συγκεκριμένο άρθρο ε, στον κανονισμό ασφαλείας των προϊόντων είναι να ενισχύσουμε την ασφάλεια των προϊόντων και να ενισχύσουμε την εποπτεία της αγοράς ώστε τα μέλη, τα μέλη να μπορούν να αναγνωρίζουν τα επικίνδυνα προϊόντα. 10% των επικίνδυνων προϊόντων όπως ανοιχθεύθηκαν από το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ε, που βρέθηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά η προέλευση δεν είναι γνωστή και 10% είναι ψηλό ποσοστό. Γι' αυτό η ένδειξη γεωγραφικής ε, προέλευσης είναι πολύ σημαντική απέτηση καθώς ε, και το όνομα του κατασκευαστού και η διεύθυνσή του. Θα πρέπει να δίδεται με έναν απλό τρόπο σε μια εύληπτη για τον καταναλωτή γλώσσα και επίσης είναι πολύ σημαντικό να το συνδέσουμε με το θέμα της εποπτείας της αγοράς γιατί ε, πρόκειται για δραστηριότητε ενίσχυση τη αγορά και είναι σημαντική και η συνεργασία με του ξένου εταίρου μα, Γιατί θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το άρθρο τη πρώτη επιτροπή αφορά όλα τα καταναλωτικά προϊόντα, είτε εισάγονται είτε όχι, ούτω ώστε να συμβατά με τους ε, εμπορικούς κανόνες. Ε, ελπίζω να είναι χρήσιμο για την επίτευξη των σκοπών αυτή τη επιτροπή και είμαι στη διάθεσή σα για την απάντηση περαιτέρω ερωτήσεων. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σπανού. Ο Σαλβατόρε Γιακολίνο είναι σκιώδες ε, εκ μέρους του ΕΛΚ και ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια συντομότατη παρέμβαση. Δεν πρόλαβα να ακούσω την ε, συγγήτρια, την κυρία Μοσκαρντίνη. Ε, αναμφίβολα πρόκειται για ένα ντοσιέ που έχει ιδιαίτερη σημασία και σαφές είναι ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να γίνει μεγαλύτερη η διασύνδεση ασφάλειας και καταναλωτών των δύο αυτών πτυχών ενός κοινού στόχου και για τα εισαγόμενα και για τα μη εισαγόμενα προϊόντα. Είναι σημαντική η έμφαση που θα δοθεί στο άρθρο 7 του κανονισμού, εκεί όπου υπήρχαν αρκετέ αμφισημίες και στο Συμβούλιο και αρκετές διαφωνίες. Και γι' αυτό είχε παγώσει ο κανονισμό για πολύ καιρό. Ακούσαμε τώρα την άποψη και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στηρίζουμε την πρόταση και θεωρούμε ότι πρόκειται για ορθή πρόταση διασφάλεια προκειμένου να βελτιωθεί η δυνατότητα επιλογή των καταναλωτών και να συσχετιστεί περισσότερο η διάσταση τη ετικετοθεσία με την εκκλασιμότητα και με συγκεκριμένε αναφορέ στι σχέσει συνεργασία με τρίτε χώρε. Εδώ βέβαια επιφυλάσσομαι να αποτιμήσω την επιλογή την δυνατότητα μάλλον να υποβάλω κάποιες μετριοπαθείς τροπολογίες που να οδεύσουν και στην κατεύθυνση των επιλογών που προέκυψαν και μέσα από την συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Κριστιανά, έχεις το λόγο για να κλείσει η συζήτηση. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, παρατηρήσεις που μας έκανε. Είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει διάθεση από την πλευρά της Επιτροπής να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε για κάτι που για μας όμως παραμένει κάπως αμφίβολο. Δηλαδή θα ζητήσουμε κάποια πράγματα, αλλά μετά μπορεί να προσκρούσουμε σε διαφορετικές επιθυμίες και απαιτήσει. Δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε εδώ τους πολίτες μας. Ευχόμαστε σε αυτή την περίπτωση το Κοινοβούλιο να εργαστεί αμελητή, προκειμένου το όλο αυτό εγχείρημα να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος της τρέχουσας θητείας. Και θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιες πτυχές που μπορούν να βελτιωθούν. Ορισμένες τις υπενήχθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις γνωρίζει. Ελπίζουμε ότι σε στα υπόλοιπα μπορεί να καταγράψει και να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις που υποβάλαμε κι εμείς στη συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ακούγοντας όσα είπαν οι συνάδελφοι, να σας θυμίσω ότι βρισκόμαστε στην αίθουσα Αλτιάς Κάσπαρη. ο οποίος ήταν ένας από τους μεγάλους εμπνευστέ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μετά τον πόλεμο. Επόμενο βήμα, επόμενα στάδια της εξέτασης του θέματος, Ιούνιο 15-16 για την εξέταση της, ε, του σχεδίου έκθεση από την τη Επόμενο σημείο στην εμερήσια διάταξη. 19. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων, συμφωνία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσική Ομοσπονδία για τι πρόδρομε ουσίε των ναρκωτικών. Είμαστε η καθήλυν υπεύθυνη επιτροπή. Ο κύριο Προύστα από το ΕΛΚ είναι ο εισηγητής μας και το δίνω το λόγο. <coughs> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία συνέψαν μια συμφωνία για τον έλεγχο και την ανταλλαγή ε, τελωνιακών πληροφοριών σε σχέση με πρόδρομες ουσίε των ναρκωτικών. Αυτή η συμφωνία η οποία θα υπογραφεί προσεχώ στην κορυφή μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, Ρωσία, στι 4 Ιουνίου στο Κατερίνενμπουργκ, είναι η τελευταία από συμφωνίε από μια σειρά συμφωνιών που έχουν συναυθεί εδώ και χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες όσον αφορά ε, το εμπόριο κάποιων χημικών προϊόντων τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν στην παρασκευή ναρκωτικών. Καθώς είμαι εισηγητής ε, για την παρακολούθηση του εμπορίου σε σχέση με αυτές τις πρόδρομες ουσίες, είμαι ιδιαίτερος ευαίσθητος ε, με το, για το θέμα αυτό και είμαι υπέρ της σύναψης αυτής της συμφωνίας. Δεν θεωρώ λοιπόν θα πρέπει να θέσουμε ένα αμφιβόλο τη σύναψη συμφωνίας του του τύπου με τη Ρωσία. Το ίδιο άλλωστε πράξαμε και με πολλές άλλες χώρες, συγκεκριμένα με τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Κίνα στο παρελθόν. Ε, σήμερα φαίνεται ότι η Ρωσία είναι μια ζώνη προορισμού ε, ε, παραπάνω από μια ζώνη τράνζιτ και διακίνησης ναρκωτικών όπως για παράδειγμα αμφεταμίνης ε, που περνάνε από την ε, Ρωσία. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστεί πιο έντονο με τη Ρωσία στη μάχη κατά των ναρκωτικών. Η συζήτηση σήμερα θα πρέπει να μα επιτρέψει να έχουμε τι αναγκαίε διευκρινήσει εκ μέρου τη Επιτροπή όσον αφορά ορισμένε πτυχέ αυτού του σχέδιου συμφωνία. Αυτό ο τύπο συμφωνία στη μάχη κατά των ναρκωτικών ολοκληρώνει την εποπτεία εμπορικών ανταλλαγών και προβλέπει ένα μηχανισμό αμοιβαία συνδρομή. Έγκυται σε μια προηγούμενη ειδοποίηση πριν από την εξαγωγή, από την εξαγωγική χώρα, ε, και ακολουθεί μια περίοδος όπου η χώρα εισαγωγής μπορεί να ασκήσει την εποπτεία στη βάση μιας ε, γραπτής δικαιολόγησης. Υπάρχει μια αμοιβαία ανταλλαγή ακόμα και εμπιστευτικών ε, δεδομένων, τα οποία είναι κατ' ουσία εμπορικά δεδομένα, αλλά μπορούν να συμπεριλάβουν και προσωπικά δεδομένα όσον αφορά το διαχειριστή μιας ε, επιχείρησης. Υπάρχουν 23 πρόδρομες ουσίες και θα πρέπει η συμφωνία να καλύπτει μια περίοδο 5 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας ε, μπορεί να ανανεωθεί αυτόματα, εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις. Ε, Ιδού λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ορισμένα θέματα και ορισμένοι προβληματισμοί για να προχωρήσει η συζήτησή μας. Η συμφωνία θα πρέπει να στηρίζεται σε ψηλό βαθμό εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών. Αλλά οι ρωσικές υπηρεσίε έχουν επικριθεί λόγω διαφθοράς και βραδιών διαδικασιών. Η Κομισιόν ε, θεωρεί ότι θα μπορέσει η Ρώσικη πλευρά να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό εφόσον μιλάμε για εμπιστευτικά δεδομένα που εξαγωγικές μας εταιρείε δεν θα ήθελα να πέσουν στα λάθος χέρια. Η Ρωσία, ωστόσο, όπως το λέει ο Ευρωπαϊκός Έλεγχος, δεν θεωρείται ως εγγύητρια επαρκούς επίπεδου προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Ρωσία δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και το πρωτόκολλο σε σχέση με την ε, εποπτεία και τις ε, διασυνοριακές ανταλλαγές δεδομένων ε, υπάρχει μια συμφωνία του 2010 μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την προστασία ταξινομημένων δεδομένων που αφορά περισσότερο πολιτικά και διπλωματικά δεδομένα παρά εμπορικά δεδομένα ε, εμπορικών επιχειρήσεων. Ε, είναι αυτό επαρκέ. Ε, επιτρέψατε μου να εκφράσω κάποιε επιφυλάξει για το θέμα αυτό, πόσο μάλλον αφού η συμφωνία δεν προβλέπει οι, τα μέρη να μπορούν να ελέγξουν την ανεξαρτησία της συμφωνίας μέρου άλλων μερών. καμία, δεν προβλέπει καμία διαδικασία ε, διακοπής, ε, μονομερούς διακοπής συμφωνίας σε περίπτωση ε, κατάφορων παραβιάσεων στον τομέα της προστασίας των εμπορικών δεδομένων. τέλος, η συμφωνία αυτή θέτει κάποια ζητήματα εμπορικής φύσεως, προβλέπει το δικαίωμα άσκησης έσταξης ε, και η Ρωσία συνεχίζει να ασκεί κάποιους ε, περιορισμούς όσον αφορά τις αγωγές γεωρικών προϊόντων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και υπεκφεύγοντας ε, στο πρόσχημα της παραβίασης υγειονομικών κανόνων εκ μέρους ορισμένων χωρών μελών. Άρα λοιπόν φαίνεται παράδοξο να γίνει μια διμερής ε, συμφωνία με την ε, Ρωσία γιατί ε, βεβαίως υπάρχουν κάποιοι τελωνακοί έλεγχοι στο, στο, στη Ρωσία, Λευκορωσία και το Καζακστάν, αλλά υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι γιατί ε, μπορεί να περάσουν οι επικίνδυνες ε, ουσίες μέσω μιας άλλης χώρας, όπως είναι η Λευκορωσία, όπου τα σύνορα είναι τροτά. Ε, θα πρέπει και οι άλλες ε, χώρες όπως είναι η Ουκρανία, η Μολδαβία να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους συμφωνίες. Ήδη λοιπόν τα είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω με ανυπομονησία τις δικές σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλει κάποιος συνάδελφος στο λόγο. Όχι. Α, ο Σαλβατόρε. Για Θα ήθελα απλά να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο εισηγητής μόλις πριν ε, για την σημασία της συνεργασίας, για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών. Γι' αυτό και τη συμφωνία αυτή πρέπει να την υποστηρίξουμε. Θα επιτρέψει ε, την ε, ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. και σε ό,τι αφορά τις ε, πρόδρομες ουσίες θα έχουμε επίσης καλύτερη δικαστική και αστυνομική συνεργασία η οποία θα δράσει στις σχέσεις εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η διάσταση αυτού του φαινομένου πλήττει πολύ και την οικονομία και σίγουρα πρέπει να στηρίξουμε τη συνεργασία αυτή. Ευχαριστώ. Thank you, Commission. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε και την Κομισιόν. Παόλο Μαζαρίνη είναι ο εκπρόσωπος. Τι έχετε να πείτε στις ε, ανησυχίες που εξέφρασε η Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Προύστ για την έκθεση σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν για την ε, σύναψη της Δημερούς Συμφωνίας με τη Ρωσία για τις πρόγραμμα των ναρκωτικών. Έχω να κάνω τα σχόλια. Πρώτα απ' όλα, τέτοιου είδου συμφωνίε σίγουρα πρέπει να βασίζονται σε σχέσει εμπιστοσύνη. Και εμεί έχουμε εμπιστοσύνη στη Ρωσική Ομοσπονδία ότι θα πράξει τα δέοντα για να εφαρμόσει τη συμφωνία. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε συμπεριλάβει κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Θα ξέρετε ότι είναι η πρώτη συμφωνία για τις πρόδρομες ουσίες των ορκωτικών που περιλαμβάνει δέσμοι διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό δεν συνέβαινε σε προηγούμενες συμφωνίες. Αν και η ανταλλαγή πληροφοριών όπως πολύ σωστά υπογραμμίσατε, εν γέννη αφορά τα εμπορικά και όχι τα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει πάντως μια δέσμη δεδομένων που ακόμη και από τον Ευρωπαίο Επόπτη για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρείται μια καλή ε, δέσμη βασικών αρχών που θα εξασφαλίσει ε, την ενδεδειγμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων και σε αυτή τη χώρα. Επίσης ε, θέσατε το ζήτημα της Τελωνικής Ένωσης. Πράγματι υπάρχει Τελωνιακή Ένωση με το Καζακστάν και τη Λευκορωσία. Το 2010 τέθηκε σε ισχύ. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησε αυτό το θέμα. Μάλλον δεν συζήτησε αυτό το θέμα στι διαπραγματεύσει ε, για τη συμφωνία για τι πρωτομουσίες ναρκωτικών. Η ρωσική πλευρά δεν θέλησε να το θίξει ουσιαστικά. Ο βασικό λόγο για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ε, να έχει διαπραγματεύσει με όλο και προτίθεται να έχει διαπραγματεύσει με όλο και περισσότερε χώρε, είναι επειδή επιθυμεί να διευρύνει αυτή την ε, συνεργασία για τον έλεγχο των προδρομονισιών. Όσο περισσότερε συμφωνίε συνάψουμε τόσο καλύτερο θα είναι ο έλεγχο. Έξω και προτείναμε και άλλες ε, συμφωνίες ε, για το μέλλον με άλλες περιφέρειες, ε, άλλες χώρες γύρω από την περιοχή αυτής της Κεντρικής Ασίας. Θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αυτό, να ξεκινήσουν δηλαδή στο μέλλον διαπραγματεύσει. Άλλες συμφωνίες που έχουμε, όπως με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, Στι περιπτώσει αυτού, το γεγονό ότι ήταν κοντά σε περιοχέ που είχαμε τέτοια διακίνηση ναρκωτικών, δεν είδαμε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα παρέκκληση με κάποιων προβλημάτων στο εμπόριο. Εν γέννη, είμαστε ικανοποιημένοι για τη στήριξη που παρέχει το Κοινοβούλιο στη συμφωνία αυτή και ελπίζουμε να ανοίξει μια νέα σελίδα ε, στην συνεργασία μας με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο σχόλιο ο εισηγητής. Μετά από άκουσε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, α, σημείωσα τις ε, προτάσεις της Επιτροπής. Πρόκειται βεβαίω για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Μπορούμε να θέσουμε το θέμα, πώς μπορούμε να δράσουμε και να ασκήσουμε πιέσεις και αν μπορεί να ανασταλεί η συμφωνία σε περιπτώσεις ε, κατάφορης παραβίασης των κανόνων για την ε, αντιμετώπιση εμπιστευτικών πληροφοριών. Άκουσα τα όσα είπε η Κομισιόν και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι συγκεκριμένο και αποτελεσματικό το ταχύτερο δυνατό γιατί στον τομέα αυτό ο χρόνος μας είναι μετρημένος. Ναι, πρόκειται για μια ε, διαδικασία ε, προβλέπεται από το Συμβούλιο, η επόμενη φάση θα είναι η εξέταση του σχεδίου έκθεσης ε, για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας στη συνάντησή μας του Ιουλίου, 10 και 11 Ιουλίου. Δηλαδή η τελευταία συνάντηση πριν από, τις, ε, από την καλοκαιρινή πάυση μου λένε ότι θα πρέπει να περάσουμε στο σημείο 24. Ε, το, 20 μάλλον. Πρόκειται μία έκθεση της ΙΤΡΕ που είναι η αρμόδια επιτροπή η συγγήτρια για, τη δική μας ε, επιτροπή είναι η Μαρία Μπαδία, στην οποία δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πριν ε, περάσω στο θέμα αυτό, θα ήθελα να ζητήσω τη δόση μας καφεΐνης. Δεν έχει προβληθεί καφέ σήμερα. Υπάρχει μια απεργία για τον καφέ. Ωραία λοιπόν. Θα περάσουμε, θα συνεχίσουμε το 24, CARS 2020. Ε, Πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα μιλήσω στα αγγλικά γιατί έχω τις σημειώσεις μου στα αγγλικά. Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά δυσχερή περίοδο με την αγορά, με μια μείωση της ε, αγοράς αυτοκινήτων για πέντε συνεχή έτη. Και αυτή η κατάσταση πιέζει πολύ τις επιχειρήσεις να διευθυνθώσουν τις δραστηριότητές τους και έχουν εξαγγείλει το κλείσιμο πολλών ε, μονάδων παραγωγής και την μείωση και απώλεια θέσεων εργασίας. Ε, υπάρχει λοιπόν μακροπρόθεσμα μία πρόκληση ούτε ώστε να βρεθούν κάποιες βιώσιμες ε, λύσεις σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να υποστηριχθεί λοιπόν η αυτοκινητοβιομηχανία στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Ε, ε υπάρχει μεγάλη ανάγκη έρευνας ε, το 2009 29 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν για την έρευνα, διότι είναι σημαντικός πολλαπλασιαστής ανάπτυξης λόγω της ε, ισχυρής διασύνδεσης με ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους. Ο κλάδος σήμερα βρίσκεται σε μια ιστορική καμπή και θα υπάρξουν σημαντικές μεταβολές σε πολλούς ε, τομείς που ούτως ώστε θα αναδιαμορφωθεί η αυτοκινητοβιομηχανία και οι αγορές παγκοσμίως. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το σχέδιο πρόγραμμα δράση. Και είναι επίσης ιδιαίτερος, ε, έρχεται η κατάλληλη στιγμή και θα πρέπει να χαιρετήσουμε αυτή την ιδέα τη επιτροπή. Καταρχήν η παραγωγή και η εμπορική εταίροι μας ε, μετακινούνται και πολλές ε, τρίτες αγορές αυξάνονται ραγδαία. Η ανταγωνιστική πίεση αυξάνεται συνεχώ και οι εταιρείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερε ε, προκλήσει στι δικέ του ε, αγορέ, ενώ αναπτύσσονται ευκαιρίε σε τρίτε αγορέ. Η ατζέντα του κλίματο επίση γίνεται όλο και πιο επιτακτική και είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί το θέμα των εκπομπών αερίων ε, θερμοκεπίου και θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματική εφαρμογή των σύγχρονων ε, τεχνολογιών σε σχέση με τις εκπομπές αερίου. Λόγω της μείωσης του εγχώριου, της εγχώριας αγοράς, το εμπόριο είναι ο μόνος, ε, η μόνη δυνατότητα ανάπτυξης. Ε, η, επιτροπή, η ανακοίνωση της Επιτροπής παρουσιάζει ένα πρόγραμμα δράσης για την αυτοκινητοβιομηχανία, το οποίο διατυπώνεται σε τέσσερις πυλώνες επένδυση σε προηγμένες τεχνολογίες και χρηματοδότηση των καινοτομιών ε, μέσω διαφόρων ρυθμιστικών πρωτοβουλειών, βελτίωση των συνθηκών της αγοράς μέσω ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά μέσω αποτελεσματικής εμπορικής πολιτικής και διεθνούς εναρμόνισης των ρυθμίσεων για τα οχήματα και προσαρμογές μέσω επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στις δεξιότητες και μειώνοντας τον αντίκτυπο της αναδιάφρωσης. Μέσω αυτής της στρατηγικής η Επιτροπή θέλει να ενισχύσει το ρόλο της αυτοκινητοβιομηχανίας και να αναστρέψει την καθοδική πορεία από το 60% ε, το ΑΕΠ στο 20% το 2020. Ε, και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Εμπορική Πολιτική θα πρέπει να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Παραγωγική Βάση και γι' αυτό όμως περισσότερο συντονισμό μεταξύ εμπορική και βιομηχανική πολιτική. Θα πρέπει επίση να μελετήσουμε προσεκτικά τι επιπτώσει των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και να ενισχύσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις γιατί έχουν ένα σωρευτικό αποτέλεσμα στην ανταγωνιστικότητα της δικής μας αυτοκινητοβιομηχανίας. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι όλα τα συμφωνηθέντα μέτρα στις συμφωνίες αυτές οικονομικών, ελεύθερων οικονομικών ανταλλαγών θα εφαρμοστούν όπως η κατάργηση των τελειωνικών διασμών. Και τέλος θα ήθελα να οργανώσω μια ανταλλαγή απόψε με τους ενδιαφερόμενους στη συνεδρία του ΙΕΝΟΥ γιατί θα πρέπει να γνωρίσουν τη δική μας θέση και εντωμεταξύ θα ήθελα να χαιρετήσω την υποβολή των δικών σα προτάσεων ε, κατά τη διαδικασία προετοιμασίας του σχεδίου γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Λοιπόν, να συζητήσουμε τώρα πρώτα απ' όλα Brent Lange από το S&D. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ Μάρια για την πολύ εξωτική παρουσίαση της ε, κατάστασης ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Πράγματι έχουμε μια δύσκολη κατάσταση και η μείωση του κέρδους ε, στην ε, Ευρώπη είναι τεράστια και έχουμε ένα υπερβολικό δυναμικό αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη Θα πρέπει να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Ε, ε, αυτό είναι το ένα. Και επίση μακροοικονομική πολιτική συνολικά, εφόσον σε πολλές χώρες της Ευρώπης υπάρχει μείωση της ζήτησης αυτοκινήτων. Και όσο και καινοτόμα να είναι η πολιτική που χαράσει κανείς, εφόσον οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν αυτοκίνητα, δεν θα το πράξουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ξεκάθαρα το μακροοικονομικό προσανατολισμό την πολιτικών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν ακριβώς στις νότιες χώρες η μείωση ε, η μείωση ζήτηση αυτοκινήτων δεν μπορεί να ενισχυθεί, δεν θα υπάρξει δυνατότητα τόνωσης της ε, αγοράς ε, εξοπλίσης του δυναμικού στην Ευρώπη. Υπάρχουν βεβαίως πολλές διαφορές στην στο επίπεδο του ανταγωνισμού. Ο ΩΣΑ έκανε μια πολύ ξεκάθαρη ανάλυση λέγοντας ότι υπάρχουν ανταγωνιστικοί και μη ανταγωνιστικοί κατασκευαστές αυτοκινήτων. Θα πρέπει νομίζω να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από τις άλλες πρακτικές των ανταγωνιστικών ε, κατασκευαστών και εδώ σημασία έχει το θέμα της καινοτομίας αλλά και της ε, συμμετοχής των ε, απασχολούμενων. Και θεωρώ ότι αυτό είναι προφανές όταν κάποιες επιχειρήσεις διαμορφώνονται μέσω του κοινωνικού διαλόγου και οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην ε, πολιτική μιας επιχείρησης και μπορούν να επιφρεάσουν ζητήματα αναδιάρθρωσης. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα την κρίση από άλλες επιχειρήσεις όπου δεν ακολουθούνται αυτές οι πρακτικές συμμετοχής των εργαζομένων. Και το τρίτο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε η Μαρία, το θέμα των εξωτερικών σχέσεων. Είναι ξεκάθαρο η ανάπτυξη, ε, βεβαίως αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα εκτός Ευρώπης, εντός της Ευρώπης, ε, στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε να διατηρήσουμε το επίπεδο των πωλήσεων. Αλλά οι επιπλέον αγορές ε, βρίσκονται εκτός της Ευρώπης και εδώ οι ρυθμίσει ε, τη δεσμεύσει με έναν των χωρών είναι απολύτω καθοριστικέ. Τρει σημαντικέ ερωτήσει. Συνήψαμε την συμφωνία, εμπορική συμφωνία με την ε, Κορέα, όπου θα πρέπει να έρθουν ε, οι, τα εμπόρια των δασμολογικά εμπόδια υπέρ των αυτοκινητοβιομηχανιών αλλά στην Κορέα υπάρχουν επιπλέον απαιτήσει για την ε, πιστοποίηση των ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Δηλαδή τα... η εισαγωγή ανταλλακτικών αυτοκινήτων προς την Κορέα δυσχεραίνεται και επιπλέον επιβάλλεται ένα επιπλέον τέλος για τα αυτοκίνητα ε, που αφορά ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Πώς προτίθεται να αντιδράσει εδώ η Επιτροπή. Και το ίδιο ισχύει και για τη Ρωσία. Βεβαίως η Ρωσία είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά και πάντοτε αντιμετωπίζουμε δυστυχώς το θέμα ότι η Ρωσία επιβάλλει ένα φόρο ανακύκλωσης μόνο για εισαγόμενα οχήματα και με τον τρόπο αυτό ε, κλείνει τη δική ε, αποκλείει την αγορά. Ε, Ευχαριστούμε πολύ η Κάθριν ε, Πύρτα από το Άλντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι αρκετά ενδιαφέρον το θέμα γιατί αφορά και τη θεώρησή μας προς το μέλλον. Δεν είναι εύκολο να κοιτάζει κανείς μια γυαλινή σφαίρα να προβλέπει τι θα συμβεί μελλοντικά. Όμως κοιτάζοντας το Εάν θέλουμε να προβλέψουμε περισσότερα ε, και να έχουμε περισσότερες σχέσεις, ίσως αυτό που να μας απασχολήσει είναι οι καλύτερες σχέσεις με περισσότερα αποτελέσματα και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις και για τις εμπορικές δραστηριότητες. Πάντοτε σκέφτομαι την ιστορία του 90 ε, και του 80 των πατεράδων στο Λονδίνο που σκέφτονταν πώς να αντιμετωπίσουν την κίνηση και το τι γινόταν με τα απόβλητα από, τα, ε, από τις άμαξες, ε, με τα άλογα, τον προηγούμενο αιώνα, τον 19ο, έπρεπε να αλλάξουν τη ζωή τους ε, σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι οι βιομηχανίες, οι αυτοκινητοβιομηχανίες συγκεκριμένα έχουν δημιουργήσει και έχουν προσφέρει τεράστια οικονομικά εφέλη στην Ευρώπη στο παρελθόν. Πάντοτε βρισκόμασταν στην πρωτοπορία των νέων τεχνολογιών. Όμως το να κοιτάζουμε διαρκώς ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες που προκύπτουν, ε, να σκεφτούμε ότι είναι, υπάρχει δυνατότητα μερικά αυτοκίνητα να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα και να εκτυπώνονται. Ή κάπως μπορεί να φτιαχτεί στο μέλλον ένα αυτόματο αυτοκίνητο που να μην χρειάζεται οδηγός για να σε πάει στο αεροδρόμιο. Πρέπει εδώ να αναγνωρίσουμε τις τεράστιες αλλαγές που προκύπτουν ε, και οφείλονται στην τεχνολογία. Εάν η Ευρώπη δεν ε, αδράξει αυτές τις ευκαιρίες και δεν αναλάβει και την ε, πατρότητα και δεν αναπτύξει τέτοιες τεχνολογίες θα μας ξεπεράσουν άλλα πιο εφάνταστα μέρη του κόσμου και με περισσότερο δημιουργικά και θα μείνουμε πίσω. Το να αναπτύξουμε λοιπόν οχήματα για την ερχόμενη 20 ετία και να στηρίξουμε την αυτοκινητοβιομηχανία με τη δική του συμμετοχή απαιτεί να ε, παρατηρούμε διαρκώς τις νέες τεχνολογίες που προκύπτουν και να μην σχεδιάζουμε μόνο με βάση το τι έχει γίνει ως τώρα, αλλά να έχουμε πάντοτε το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον. Πρόεδρος, ο κύριος Μέρφυ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι τεράστιο το θέμα. Πρόσφατα ο κύριος Μαρκιόνε προέβλεπε μια άσχημη τροπή για την αυτοκινητοβιομηχανία και όντως ε, υπάρχει θέμα με τις υπερβολικές δυνατότητες παραγωγής που ήδη υπάρχουν. Ποιος θα αντιμετωπίσει εδώ τον κίνδυνο είναι το ερώτημα. Η άποψή μου είναι ότι οι εργαζόμενοι θα την πληρώσουν. Οι εργαζόμενοι στις αυτοκινητοβιομηχανίες, διότι η κλίμακα της κατάρρευσης της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστια. Από 17 εκατομμύρια το 2012 έχουν πουληθεί πλέον 12,5 εκατομμύρια οχήματα. Και αυτό δείχνει πόσοι πολίτες αλλάζουν την σχέση τους ε, με το αυτοκίνητο. Και ούτω ή άλλω υπήρχε υπερβολική παραγωγή στην Ευρώπη πριν την κρίση. Υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια στην Ευρώπη. Πολλοί κατασκευαστές χάνουν χίλια ευρώ ανά αυτοκίνητο την ημέρα στις πωλήσει του λόγω της υπερβολική δυνατότητας και το ερώτημα είναι ποιο θα καταβάλει το τίμημα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μηχανία μα. Θα πρέπει να κοιτάξει από την άποψη τη αναδιάρθρωση το τι έγινε στι ΗΠΑ. Όμω σκεφτείτε τι έγινε εκεί ακριβώ. Ε, μια τεράστια αναδιάρθρωση με αποτέλεσμα να ε, καταστραφεί εν μέρη κάτι που ήταν καλοπληρωμένη θέση εργασίας. Οι καλοπληρωμένες αυτές σταθερές θέσεις εργασίας χάθηκαν. Έγιναν ε, χαμηλής αμοιβής θέσεις με μικρή προστασία από συνδικαλιστές οργανώσεις και είναι σαφές ότι και για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές εάν ακολουθήσουν αυτή την πορεία θα υπάρξει αντίσταση. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αντισταθούν, διότι θα πληρώσουν τα σπασμένα οι εργαζόμενοι για τις απώλειες των αυτοκινητοβιομηχανιών. Αντιστροφή των πολιτικών λιτότητα χρειάζεται, κατά τη δική μου άποψη, αλλά και αναδιάρθρωση τη αυτοκινητοβιομηχανία γενικά. Η ανακοίνωση λοιπόν είναι μια απόπειρα να αρθρώσει κάτι τέτοιο, αλλά δεν βλέπω να είναι συνεπής η προσέγγιση. Διότι το σύστημα με ξεχωριστή ιδιοκτησία των βασικών αυτοκινητοβιομηχανιών, ο ανταγωνισμός μεταξύ τους, ενώ κάποιες τα πηγαίνουν σχετικά καλά ακόμα, όπως η Volkswagen, ενώ άλλοι η Fiat, η Peugeot αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα σε εξατομικευμένη βάση να αναδιορθωθεί η, η παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Και θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Κατά την άποψή μου λοιπόν δεν περιμένω να φτάσει σε εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά αυτό που προτείνατε θα έπρεπε να οδηγήσει σε δημόσια ε, ανάληψη της ε, ευθύνης, να υπάρξει πράσινη κινητικότητα ή να υπάρξει επένδυση στην μετατροπή της παραγωγής σε άλλες κοινωνικώς χρήσιμες ε, μορφές όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες και εκεί να στραφεί η αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό είναι που, χρειαζόμαστε και έτσι θα μπορούσαν να σωθούν οι θέσει χρειαζομαστε και ετσι θα μπορουσαν να σωθουν οι θεσεις εργασια Και προ όφελο των αυτοκινητοβιομηχανιών. Οι επικεφαλείς θα μπορούσαν να προστατεύσουν έτσι και το κέρδος τους ε, με κάθε κόστος αντί να πλήξουν του εργαζομένου. Θα Έχουμε σοβαρούς αγώνες και μάχες σε πολλές χώρες της Ευρώπης, νομίζω, γιατί οι εργαζόμενοι στις αυτοκινητομηχανίες θα κάνουν το παν για να προστατεύσουν τις δικές τους θέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλες παρεμβάσεις. Να σας πω, σε ό,τι αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, δεν πρέπει να παραλείπουμε και τις απόψεις όσων έρχονται από τη Γαλλία και την Ιταλία. Είναι χώρες με παράδοση στο χώρο, αλλά δεν θέλω να τοποθετηθώ εγώ εκ μέρου του Ας ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη φορά ο κύριος Φιλίπ Ζων από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να, πούμε, να πω, παρότι περιμένουμε με αδημονία την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής σας για πολλαπλούς λόγους. Ιδιαιτέρως γιατί η διεθνής διάσταση ε, λαμβάνει όλο και περισσότερη σημασία για την αυτοκινητοβιομηχανία διότι όταν σε αυτό το πρόγραμμα δράση, την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, ε, μιλάμε για αυτό τον τομέα, δεν μιλάμε μόνο για του παραγωγού αυτοκινήτων, αλλά για το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αλυσίδα. Την παραγωγή, τα ανταλλακτικά, τη διανομή και ούτω καθεξή, όπω είπε ο εισηγητή. Οι διεθνεί πτυχέ ε, λαμβάνουν μεγαλύτερη σημασία και βάρο, ακριβώ γιατί βρίσκεται σε τέλμα η ευρωπαϊκή αγορά. Ε, Μα ενδιαφέρει περισσότερο η αγορά των τρίτων χωρών, γιατί εκεί υπάρχουν περισσότερε δυνατότητε ανάπτυξη. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι θα μπορούσε να έχει μέλλον η αυτοκινητοβιομηχανία αρκεί να εξοπλιστεί, να θωρακιστεί για να παράγει προϊόντα τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη και τις ανάγκες των τρίτων χωρών. Στρατηγικές λοιπόν για εμπορικούς ε, σκοπούς και έπειτα Ω τώρα η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές εταιρείε ήταν στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει ρήξη και να μην ε, συνεχίζεται αυτή η θετική πορεία. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν από την άποψη της έρευνας ή από τη ρύθμιση για την ασφάλεια, για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο το επίπεδο του το διαγνωστικό, αλλά και της προσπάθειας εναρμόνισης των ρυθμίσεων. Έχουμε εντατικές διαπραγματεύσεις με τους μεγαλύτερους εμπορικούς μας εταίρους ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Ε, δέχομαι λοιπόν εδώ με μεγάλη χαρά την πρόταση του εισηγητή να οργανωθεί εργαστήριο τον Ιούνιο για τα θέματα αυτά. Είμαστε στη διάθεση και της Επιτροπής σας και του εισηγητού σας για να δώσουμε κάθε ε, χρήσιμη συνεισφορά στη συζήτηση αυτή γιατί είναι σημαντικό το ζήτημα. Συνέπεια μεταξύ βιομηχανικών, εμπορικών πολιτικών και ρυθμιστική προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ωραία. Έχετε κάποια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, ίσως θα μπορούσε να μας πει κάποια πράγματα ε, για το εμπόριο με την ε, Κορέα, τη συμφωνία με την Κορέα και τους εμπορικούς φραγμούς. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάγκα έχει απολύτως δίκιο. Υπάρχει μια ε, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Κορέα που δεν αφορά το θέμα των τελωνιακών δασμών αλλά τη δυνατότητα να υπάρξουν κοινέ προδιαγραφές που μπορούν να γίνουν αποδεκτές ή να γίνονται σεβαστές όταν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας όσον αφορά την νομοθεσία για τις εκπομπές αερίου ή για τις προδιαγραφές ασφάλειας να εφαρμόζονται. Και εξετάζουμε ένα παράρτημα για αυτές τις τεχνικές ρυθμίσεις, κάτι το οποίο είναι δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά θέλουμε να έχουμε κάποιους κοινού κανόνες, κοινέ ε, ρυθμίσεις ε, που θα εφαρμοστούν από την Κορέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να ελαχιστοποιηθούν, να μειωθούν τα, μη ε, τα, τα, τα εμπόδια που δεν αφορούν τους τελωνιακούς δασμούς το κείμενο εδώ δεν καλύπτει όλες τις ε, διατάξεις, ε, καλύπτει περίπου το 1 τρίτο των διατάξεων και υπάρχει ένα πεδίο όπου δεν μπορούμε να βρούμε κοινέ ε, προδιαγραφές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας. Για παράδειγμα, σχετικά αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, τι μπορεί εδώ, εξετάζω τι μπορεί να γίνει συμπληρωματικά εκ μέρους της Κορέα και ιδιαίτερα σαν αφορά τα ταλλακτικά αυτοκινήτων. Ε, άρα έχει δίκιο ο κ. Λάγκε, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Η Κορέα προτίθεται να αναλάβει κάποιες νέες πρωτοβουλίες νομοθεσίες ε, που για την ε, Κορέα αντιβαίνουν το πνεύμα της συμφωνίας που λέει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν επιπρόσθετες διατάξεις αλλά εμείς από την πλευρά μας έχουμε κάποιες δυσκολίες όσον αφορά ορισμένα επιπλέον μέτρα όπως αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Λάγκε. Αλλά μπορούμε να πούμε στον κύριο Λάγκε, οι συνάδελφοι που είναι υπεύθυνοι ε, για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων ε, υπό την εποπτεία του Επιτρόπου Ντεχούχτ, ασχολούνται με τα θέματα αυτά και οι διατάξεις ανταλλακτικά αντιβαίνουν με το πνεύμα των συμφωνιών πράγματι που λέει ότι δεν θα πρέπει να θεσπιστούν νέες ε, απαιτήσει. Εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της ε, Κορέα. Η Μαρία έχει το λόγο για να κάνει κάποια τελικά σχόλια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας θα έλεγα ότι συμμερίζομαι τα όσα είπατε και θα ήθελα απλώς να παρατηρήσω ότι βεβαίως ε, χαίρομαι που συμφωνείτε μαζί μου ότι αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο θέμα εδώ που αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία και την οικονομική κατάσταση στις αστικές περιοχές, τη σημασία της εξωτερικής αγοράς, των εξωτερικών αγορών, να δώσουν μια απάντηση σε αυτή την κατάσταση, επίσης τη σημασία των καινοτομιών και τη δυνατότητα να είμαστε ξεκάθαρες προς το είδος των καινοτομιών που επιθυμούμε, γιατί όπως είπε ο εκπρόσωπος του Άλντε, θα πρέπει να βελτιώσουμε την ε, δική μας παραγωγή, αλλά εστιασμένη προς το μέλλον ε, και βεβαίως σε σχέση με τους ε, κινδύνους που ενέχουν οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών θα πρέπει να δούμε πολύ συνειδητά της υποεξέλιξης συμφωνίες ή τις μελλοντικές ε, συμφωνίες ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι κοινοί κανόνες και οι κοινέ προδιαγραφές αλλιώς θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει αμοιβαιότητα στην αγορά αυτή. Και σε σχέση με τα όσα είπε ο Πολ Μάρφη, πραγματικά συμμερίζομαι τις ανησυχίες του. Βεβαίως ε, όταν είπε ότι το τμήμα του προβλήματος είναι η υπερβολική ενίσχυση των μέτρων ε, λιτότητας, ε, εδώ συμφωνούμε απολύτως, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε κάποιες απαντήσεις για το ε, απολύτως εγγύς μέλλον, καθώς και απαντήσεις για το απότερο μέλλον. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να βρούμε αυτές τις απαντήσεις, γιατί ο κλάδος νοσεί ε, οι θέσει απασχόληση συρρυκνώνονται. Χρειαζόμαστε κάποιε απαντήσει. Θα πρέπει να είμαστε αρκετά έξυπνοι, τους, ώστε να σχεδιάσουμε και το μέλλον του κλάδου. Ε, σας ευχαριστώ και πάλι για όλα τα σχόλιά σας και ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ξανά για το θέμα αυτό στη βάση των τροπολογιών κλπ χρονοδιάγραμμα για το θέμα αυτό. Χθε εγκρίθηκε από του συντονιστέ. Η δεύτερη ανταλλαγή απόψε θα γίνει τον Ιούνιο σε τακτική συνεδρίαση, εξέταση του σχεδίου έκθεσης τον Ιούλιο και ψηφοφορία τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το τέλος του σημείου 24. Μετά θα συζητήσουμε με τον Επίτροπο Ντέχου, το οποίο όμως ακόμη δεν έχει φτάσει. Έρχεται σε 6-7 λεπτά. Προτείνω λοιπόν ένα σύντομο διάλειμμα. Νομίζω ότι καφές προσφέρεται εκτός της αίθουσα. Δεν ε, είναι ο καταπληκτικότερος, αλλά παρακαλώ εκμεταλλευτείτε το διάλειμμα για να πάτε ως εκεί και όχι μακρύτερα. Εγώ αυτό θα κάνω. Ευχαριστώ.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 maybe in the uh, end Την προσοχή σας παρακαλώ. Let's uh, our Να συνεχίσουμε με το σημείο 21, δηλαδή ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Ντέχου σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2013 και 2014 στα πλαίσια του επανομαζόμενου διαρθρωμένου διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέταρτος γύρος ε, διαλόγου. Και πλησιάζουμε στο τέλος και των δυο μας, της θητείας μας δηλαδή. Σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα. Γι' αυτό λοιπόν, μέλη της Επιτροπής, σας ενθαρρύνω να παρακολουθήσετε με προσοχή τη συζήτηση αυτή. Όχι μόνο γιατί μπορεί να έχετε την ε, ε, βλέψη να παραμείνετε μέλη της επόμενης θητείας, αλλά για να ξέρουμε και τι κάνουμε. Κύριε Δεχούχτε, καλώς ήρθατε και πάλι, έχετε το λόγο. Thank you. Ε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Η θητεία μου δεν λύγει την 31η Μαΐου. Οπότε πρέπει να παραμείνω μέχρι την 1η Οκτωβρίου στη θέση μου. Αν έχουν ολοκληρωθεί βέβαια όλες οι ακροάσεις ε, μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Μάλλον ε, θα βρω έναν σύμμαχο στο επόμενο κοινοβούλιο. Τέλος πάντων, να μην λήξει η ιστορία όλη αυτή την 1η Νοεμβρίου, τέλος πάντων. Σίγουρα υπάρχει ένα τέλος σε όλα. Έτσι είναι τα πράγματα. Ας ξεκινήσω λοιπόν ευχαριστώντας ε, για την πρόσκληση σε αυτόν τον τακτικό διαρθρωμένο διάλογο. Σε ένα χρόνο λίγη η του Κοινοβουλίου και σε 1,5 λιγότερο ε, λίγη θητή της Κομισιόν αλλά παρόλα αυτά εμείς είμαστε ακόμη προσιλωμένοι στα νομοθετικά μας καθήκοντα. Είναι λοιπόν πολύ νωρίς ε, να κάνουμε τον απολογισμό μας γιατί έχουμε ακόμη μέλλον μπροστά μας. Τούτου λεχθέντος, ε, ο στόχος του διαρθρωμένου διάλογου είναι σίγουρα να περνέσουμε κάποια επιτεύγματα και εγώ θα αναφερθώ σε τρία ζητήματα. Το Δεκέμβριο είναι το Συμβούλιο της Συμφωνίας με Κολομβία, Πέρου και Κεντρική Αμερική. Από την 1η Μαρτίου φέτος ε, εφαρμόζουμε με το Περού την ε, συμφωνία, ενώ για τους άλλους δύο εταίρους οι χώρες αυτές ε, ολοκληρώνουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες και ελπίζουμε για την Κολομβία να μπορούμε να εφαρμόσουμε προσωρινά τη συμφωνία από 1η Ιουλίου. Εκτός από την Γουατεμάλα, όλες οι χώρες Κεντρικής Αμερικής ε, είναι πεπισμένες ότι μπορούν μέχρι τις 15 Ιουλίου να έχουν εφαρμόσει την συμφωνία τους προσωρινά μάλλον να έχουν κάνει όλες τις ε, διατυπώσεις ώστε να μπορούμε μετά το φθινόπωρο να εγκρίνουμε ε, την προσωρινή εφαρμογή. Έχει γίνει σκληρή δουλειά, ήταν επιτυχημένες ε, οι προσπάθειες, θα στηρίζουμε τις εμπορικές συμφωνίες θέλοντας να έχουμε την αηφόρο ανάπτυξη. Πολλές φορές Έχουμε αντιμετωπίσει και κάποιε προκλήσει. Ξέρουμε τι έγινε με τη Γερμανία πρόσφατα, αλλά προσπαθούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα. Ακούμε τώρα ότι η δημόσια συζήτηση για τι δύο αυτέ συμφωνίε στα Εθνικά Κοινοβούλια δεν ήταν τόσο εντατική όσο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Σας ε, παρακαλώ λοιπόν ε, από τις εκλογικές σας περιφέρειες και με τις σχέσεις που έχετε ε, στις χώρες σας να βοηθήσετε να στηριχθεί το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης πριν από ένα χρόνο εγκρίναμε την ε, μεταρρύθμιση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Χάρη στη δική σας στήριξη είναι πιο δίκαιο πλέον το σύστημα, λειτουργεί, είναι ένα από τα πλέον γενναιόδωρα, να μην πω το πιο γενναιόδωρο από τα ισχύοντα συστήματα γενικευμένων προτιμήσεων της προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Χαιρετίζω λοιπόν και την, προηγούμενη, ε, την ψηφοφορία της προηγούμενης εβδομάδας ε, για την επέκταση του συστήματος ε, στη Μιανμάρ, ε, Βιρμανία, κάτι που δεν ήταν προβλεπόμενο όταν είχαμε εγκρίνει την πρότασή μας το Μάιο του 2011. Επεξεργαζόμαστε τώρα στην Κομισιόν ε, μία δέσμη κατεξοδότηση πράξεων για τους νέους κανόνες και πάλι εδώ θα είναι αποφασιστική στήριξή σας. Τέλος, ε, οι εμπορικές μας σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ, τροποποίηση του κανονισμού πρόσβαση στην αγορά ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη σχέση μας με τους ε, εταίρους αυτούς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοδομητική σας στάση απέναντι στο θέμα αυτό, ιδίως να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πρόκειται για μια απόφαση που θα ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να συνάψουμε τις, ε, για να μάλλον να ολοκληρώσουμε τις περιφερειακές μας διαπραγματεύσεις και να έχουμε μια πιο μακροχρόνια σχέση. Μπορούν πλέον όλες οι συμβαλόμενες πλευρές να αποφασίσουν για το τι είδους ε, εμπορική σχέση θέλουμε να έχουμε αφού πλέον όλες οι πλευρές έχουν εκφράσει ε, τις απόψεις τους. Θα έχω και μια, ε, ένα ταξίδι στην περιοχή, ε, ένα στην Αφρική συγκεκριμένα, ένα το καλοκαίρι και ένα το φθινόπορο. Σίγουρα θα λαμβάνουμε βέβαια υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις. Πάντως πρόκειται για σημαντικές αποφάσεις Έχουμε και άλλες βέβαια νομοθετικές ε, προτάσεις ε, επιτάπητος. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας από αυτών των θεμάτων προτού διακόψει το κοινοβούλιο εργασίες. Το πριν από δύο μήνες είχα κάνει και μια πρόταση για εξυγχρονισμό ε, των ε, εμπορικών αμυντικών μηχανισμών. Θα ήθελα να έχουμε ολοκληρώσει μέσα στην ε, περίοδο αυτή τις εργασίες μας για να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς εμπορικούς μας εταίρους ότι τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές δεν θα τις ανεχθούμε. Θέλουμε να έχουμε παντού θεμητό ανταγωνισμό. Νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη ευκαιρία στα χέρια μας και δεν πρέπει να τη χάσουμε. Βέβαια για να γίνει αυτό θα πρέπει να αλλάξει η ισορροπία των εμπορικών αμυντικών μηχανισμών. Είναι οι πιο προηγμένοι αυτοί οι μηχανισμοί. Προτείνουμε λοιπόν ένα δίκαιο ισορροπημένο πακέτο μέτρων που θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα αυτών των μέσων. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτες για την πρόταση αυτή. Εμείς Είμαστε αποφασισμένοι από την πλευρά της Κομισιόν να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, για να έχουμε εμπόριο δίκαιο ε, απέναντι σε όλους μας τους ε, σημαντικούς εμπορικούς εταίρους. Ένα άλλο θέμα που εκκρεμεί είναι η χρηματοοικονομική ευθύνη σε ό,τι αφορά την επίλυση εμπορικών διαφορών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σημερίζεται σε μεγάλο βαθμό την προσέγγισή μας και με ικανοποιεί αυτό, αλλά πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι το Συμβούλιο τίνει προσθέσεις ε, που θα αποτρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από το να μιλά με μια φωνή στο διεθνή ε, στίβο. Αυτό ε, έχει ως κίνδυνο την διατάραξη της διεθνούς ισορροπίας και την μη ικανοποιητική πράσπιση των ευρωπαϊκών συμφέροντων. Θα είμαστε αντίθετοι λοιπόν στις ιδέες αυτές και ελπίζω να μας στηρίξει το Κοινοβούλιο η Ολομέλεια ε, ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό μας ενθαρρύνει. Επίσης, βασιζόμαστε στη στήριξή σας ε, σε ό,τι αφορά την πρόταση για ένα διεθνές μέσο προμηθειών, δημοσίων συμβάσεων. Είναι ένα λεπτό ζήτημα η πρόοδο που σημειώνεται στο Συμβούλιο είναι πολύ αργή. Παρ' όλα αυτά θέλουμε και εδώ να δείξουμε ότι η εμπορική μα ε, πολιτική είναι αποφασιστική. Στηρίζουμε ε, λοιπόν τι ελπίδε μα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συζητήσουμε μαζί και τι προτάσει ε, που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτίωση του μέσου αυτού. Περιμένουμε λοιπόν και την έκθεση του Κοινοβούλου. Τέλο, ο κανονισμό επιβολή ομοθεσία είναι ένα άλλο κομμάτι του πάζλ που θα εξασφαλίσει ότι μπορεί αποτελεσματικά η Ένωση να να προασπίσει τα συμφέροντά τη και ελπίζουμε να τεθεί σύντομα σε ισχύ ώστε να ολοκληρωθεί και το θέμα αυτό στη διάρκεια αυτή τη κοινοβουλευτική περίοδου. Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τι ε, ε, διαπραγματεύσει ε, που έχει αναλάβει σε επόμενε εβδομάδε. σε επόμενου μήνε. Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις μετέρους όπω είναι η Ιαπωνία, η Ινδία, το Μαρόκο, η Ταϊλάνδη και θα ολοκληρώσουμε τις συνδιαπραγματεύσεις με τον Καναδά, την Αρμενία, την Γεωργία και τη Μολδαβία. Ελπίζω τον Ιούλιο να είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Εν συντομία θα ήθελα να μιλήσω για την ε, συμφωνία, μάλλον για την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα σε ό,τι αφορά την κατάργηση ρυθμιστικών δασμολογικών εμποδίων σε αυτή τη διατλαντική αγορά, τη διευρυμένη, νομίζω θα είναι προ όφελο όλων των ε, πλευρών, ε, των οικονομιών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των ΗΠΑ. δούμε και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οικονομίε μα ε, σήμερα, μπορεί ε, ίσως να μην συμφωνούμε με την ανεξάρτητη μελέτη που τονίζει τα ωφέλη αυτά, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι διατλαντικό εμπόριο, επενδύσεις αν δεν έχουμε ε, μία ε, συμφωνία ε, TTIP δυναμική, δεν θα τα πετύχουμε. Ζητά με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο να έχουμε μία διαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών που θα γίνει σε βάθος, θα είναι αναλυτική, διεξοδική για να εξασφαλίσουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη. Σε ό,τι αφορά την εξαίρεση του οπτικοακουστικού τομέα, λυπούμε γι' αυτό, αλλά δεν έχει τελειώσει το ταξίδι μας, καθώς πρέπει να λάβει απόφαση και το Συμβούλιο από αυτού. Εμείς πάντως θα θέλαμε να είχαμε την πιο διαβριμένη εντολή ε, την πιο διευμένη δυνατή εντολή, γιατί αν έχουμε μια περιοριστική εντολή δεν θα δώσουμε ε, στο TTIP το εύρος που απαιτείται. Και βέβαια έχουμε υπόψη μα όχι μόνο τη διατλαντική οικονομία αλλά και το παγκόσμιο εμπόριο. Γιατί η Επιτροπή ΙΝΤΑ θα είναι στο επίκεντρο μια ε, πραγματικά μάχη συμφερόντων όταν ξεκινήσουν ε, πραγματικά οι διαπραγματεύσει. Διότι την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε κάποια συμφέροντα που δεν ήταν τόσο ορτά, ε, ναυτιλία, γεωργία, υπηρεσίες, οπτικός γεωγραφικέ γεωγραφικές ενδείξεις, αέριο και άλλοι τομεί σημαντικοί της διατλαντικής οικονομίας. Αυτά όλα τα θέματα θα ανακύψουν και γι' αυτό θέλω ε, να επιτρέψετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη και στο ψήφισμά σας να δώσουμε πιο φιλόδοξα αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις. Έρχομαι τώρα στο πολυμερές μέτωπο. Περιμένουμε το Κοινοβούλιο να στηρίξει και όχι να υπονομεύσει τις προσπάθειες που καταβάλουμε ώστε στην Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕΤΟ, και Δεκέμβριο στον Παλί να μπορούμε να έχουμε ένα πολύ σημαντικό πακέτο μέτρων για τη διευκόλυνση, την εμπορική διευκόλυνση και επίσης ε, θα συνεργαστούμε και με άλλα μέλη του ΠΟΕ για μια συμφωνία εμπορίου ε, στον τομέα των υπηρεσιών. Προτείνουμε επίσης το Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Κίνα Αναμφιβολά το παγκόσμιο εμπόριο είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που θα βγάλει από τη φτώχεια εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε όμως ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο υπεύθυνη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού. Ιδίως όταν βλέπουμε να χάνονται ζωές λόγω των αποτροπιαστικών συνθήκων εργασία. Θα πρέπει να αναπτύξουμε δυνατότητες ε, εκεί που καταστρέφονται από τις εμπόλεμες συγκρούσεις που σώπουν σε κάποιες περιοχές. Τα πρόσφατα γεγονότα στο Μπαγκλαντές επίσης ε, πραγματικά ε, άγγιξαν μια πολύ ευαίσθητη χορδή εδώ στην Ευρώπη και πραγματικά μας ανησυχεί ιδιαίτερα η ασφάλεια, οι συνθήκες εργασίας σε ορισμένες βιομηχανίες, στον Παγκλαντές ή σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Αναφέρομαι και στις ε, πράξεις ε, ε, και τις ενέργειες παρακολούθησης από πλευρά της Κομισιόν. Σας εξέθεσα την προηγούμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια. Θέλουμε να έχουμε μια υπεύθυνη διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού. Μετά τη συνάντησή μας θα συναντηθώ εδώ στις Βρυξέλλες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαγκλατές για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερο πέργασιακο περιβάλλον, ποιε είναι οι προτεραιότητές μας εκεί. Θέλουμε ε, να έχουμε τη συνεργασία και των ΗΠΑ προς τον τομέα αυτό. Επίσης, ε, στο πλαίσιο του Διεθνές Γραφείου Εργασίας και με τη ΣΥΠΑ και με τον Μπαγκλαντές εργαζόμαστε για να έχουμε μια συνάντηση των εμπλεκομένων φορέων στις αρχές του Ιουλίου για να έχουμε δράσει που θα στηρίξουν το έργο που έχει ήδη ξεκινήσει μετά από αυτές τις τραγωδίες. Φυσικά θα σας στηρίσουμε ενήμερους για τις μελλοντικέ εξελίξεις στο μέτωπο αυτό. Η υπεύθυνη διαχείριση της αλυσίδας εφοδισμούς αφορά βέβαια και το τομέα της μεταπής αλλά και ε, τον εξοριστικό, εξορυκτικό τομέα. Η διαφάνεια είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για να έχουμε θετικές εξελίξεις σε χώρες που είναι ε, πλούσιες ε, σε πρωτοπαραγωγικούς ε, πόρους. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε και μια πρωτοβουλία για τα μεταλλεύματα τα οποία προέρχονται από περιοχές υψηλού κινδύνου ή που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση θα μπορούσαμε να δούμε αν θα μπορούσαμε να έχουμε λοιπόν για τη διαφάνεια ε, της αλυσίδας ευωδιασμού, για τη δέουσα επιμέλεια, στις εξωτικές δραστηριότητες, θα μπορούσαμε να έχουμε μια πρωτοβουλία, ένα σχέδιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσωπικά θα κάνω πάντο δυνατόν για να ξεκινήσουμε και μια νομοθετική πρωτοβουλία για το θέμα αυτό πριν το τέλος ε, του έτους. που φαίνεται είναι και η προθεσμία, η λήξη προθεσμία για την ε, υποβολή νομοθετικών προτάσεων. Ολοκληρώνοντα, ε, δεν επαναπαυόμαστε στι δάφνε μα και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα, όπω σα είπα και πριν, ίσω και με νέε πρωτοβουλίε πιθανόν. Βασίζομαι στη ε, δική σα προσήλωση και δέσμευση και είμαι και βέβαιος ότι θα κάνετε κι εσείς ό,τι μπορείτε για να ολοκληρώσετε τις δικές σας εργασίες και από πλευρά σας μπορείτε να βασίζεστε σε μένα ότι για το υπόλοιπο της θητείας μου θα κάνω πάντο δυνατόν ώστε να προχωρήσουμε σε διάφορα ζητήματα. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πέτρο Πεντεχούχ. Θα ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτησή μας. Η Επιτροπή επικέντρωσε την προσοχή της σωστά σε ό,τι απομένει να γίνει μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου ε, και τώρα θα, πάρουν, θα πάρετε εσείς το λόγο θα σεβαστούμε την ιεραρχία των πολιτικών ομάδων ανάλογα με το μέγεθός τους θα ξεκινήσει ο κύριος Γκασπάρη από το ΕΛΚ. Αξάτιμα κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε πολύ που σήμερα και πάλι προσήλθατε εδώ και νομίζω ότι σωστά επισημαίνετε ορισμένες επιτυχίες τις οποίες ε, χρωστάμε στην κοινή μας ε, συνεργασία τελευταία τρία χρόνια, ιδιαίτερο την προγραμματισμένη συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ελπίζω τον ε, Ιούνιο τελικά να υπάρξει οριστική συμφωνία. Είναι κάτι το οποίο δεν αναμέναμε εδώ στο Κοινοβούλιο και θα χαιρόμουν αν εσείς ε, προσπαθούσατε να κινητοποιήσετε επαρκείς ε, πόρους στην Κομισιόν, ούτω ώστε οι διαπραγματεύσεις αυτές να μπορούν να γίνουν ε, εντατικά και αποτελεσματικά, γιατί υπάρχουν πολλές διαπραγματεύσει που εκκρεμούν εδώ και χρόνια και δεν εξελίσσονται σωστά. Γιατί νομίζω ότι όσον αφορά αυτή τη συμφωνία, ε, η οποία είναι στρατηγική σημασία, θα πρέπει να επενδύσουμε όλες μας τις δυνάμεις, ούτω ώστε να μην ε, γίνει μια τέρμονη ιστορία, αλλά να οδηγηθούμε σε αυτά αποτελέσματα. Αναφερθήκατε στην, ε, στην Συμφωνία Προστασίας των Επενδύσεων με την Κίνα ε, δεύτερον, ε, είναι σημαντικό να εργαστούμε γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Κίνα και θεωρώ ότι θα πρέπει να επενδύσουμε τι προσπάθειέ μα, ούτω ώστε να βελτιωθούν οι επενδύσει μα στην Κίνα. Όταν μιλάμε όμω για προστασία επενδύσεων, η εντύπωσή μου δεν είναι ότι μόνο η Επιτροπή ε, θέλει να κάνει μια νέα συμφωνία ε, για την προστασία των παιδιών στην Κίνα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ε, χώρες που θέλουν δημερώς να συνάψουν τέτοιες συμφωνίες. Μέσα στη διαδικασία της υποτροπολογίας είχαμε 10, 15 ή 20 τέτοιου είδους ε, σχέδια ε, για διμερείς ε, συμφωνίες προστασίας των επενδύσεων. Εμείς θέλουμε να διαπραγματευτούμε τώρα με το Βιετνάμ για σύναψη εμπορικής συμφωνίας και παρόλα αυτά μια χώρα μέλος ζήτησε και, και έλαβε την έγκριση να κάνει μια διμερή συμφωνία με το Βιετνάμ. Το ερώτημά μου έχει ως εξής. Ε, Πώ θέλουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα εδώ, δηλαδή ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα για την σύναψη συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων και από την άλλη, κατά την άποψή μου, όλο και περισσότερο οι χώρε μέλη αρχίζουν να διαπραγματεύονται δικέ του συμφωνίε προστασία των επενδύσεων. Θέλετε, ε, ε θεωρείτε δυνατό να επιστήσουμε την ε, προσοχή των χωρών μελών σε αυτό το πρόβλημα, ώστε να είναι πιο συνετά τα κράτη-μέλη. Ε, δεύτερον, έχω την εντύπωση ότι κατά τον οικονομικό σχεδιοσμό δεν αναδιανέμουμε τους πόρους εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δούμε όλα τα project τα οποία σχεγραφίστε σήμερα, ε, τα οποία θέλετε να τα υλοποιήσετε με το δικό σας επιτελείο, ε, εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις και το συγκεκριμένο μου ερώτημα είναι πώς ε, μπορούμε εμείς να σας βοηθήσουμε από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια είδους διάθεση, τουλάχιστον στη δική μου πολιτική ομάδα, να σας βοηθήσουμε ούτω ώστε να υπάρξουν περισσότεροι πόροι από τις λιγότερο φορτωμένες γενικές διευθύνσεις ούτως ώστε να διοχετευθούν οι πόροι στην ε, δική σας, ε, ε, για σας, για το δικό σας έργο, το οποίο είναι πολύ πιο επαχθές. Άλλο θέμα, υπάρχει μια πλατεία συζήτηση όσον αφορά τη διαδικασία αντι-dumping για, τα, για τις ηλιακές εγκαταστάσεις. Ε, και εδώ αναφέρονται ποσοστά μέχρι το 74%. Ε, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτά τα ποσοστά, αλλά όταν αναφέρεται ένας τέτοιο ρυθμός, 47% ε, συγγνώμη, ή κατά πόσο είναι δεδειγμένο το 60% ή το 30%. Αλλά σας ελπίζω ε, παρακαλώ, γιατί δεν είναι δυνατόν εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να ενδώσουμε. Δεν είναι δυνατόν πολλές ε, χώρες ε, μέλη να πιέζονται από τους φίλους μας στην Κίνα. Θα ήμουν ευγνώμων εάν πράτατε αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε δηλαδή να επιβάλλετε τους προσωρινούς δασμούς εάν εφαρμοστεί αυτό το οποίο έχει προβλεφθεί και αν υπάρξει πίεση να συστήσουμε με τους Κινέζους, γνωρίζουμε από το παρελθόν πόσο δύσκολο είναι να διαπραγματευτούμε ένα τόσο μεγάλο εταίρο όπως είναι η Κίνα. Αλλά νομίζω ότι αν ενδώσουμε εδώ, αυτό θα επιδεινώσει τη δική μας κατάσταση. Και στη δική μας Επιτροπή Εμπορίου κανείς δεν επιθυμεί έναν εμπορικό πόλεμο με την Κίνα. Ε, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι δεδειγμένο αλλά νομίζω ότι ένα περιθώριο αντι-dumping 47% ε, είναι σημαντικό να σκεφτούμε, να εξετάσουμε τη λήψη κάποιων αμυντικών ε, μέτρων και θα σήμουν ευγνώμων εάν πραγματικά δεν ενδώσετε στο θέμα αυτό και επιβάλλετε τα προσωρινά, τους προσωριανούς ε, τελωνιακούς δασμούς που έχουν προβλεφθεί γιατί ε, η περίπτωση της Κίνας είναι συμπτωματική όσον αφορά τη διαδικασια αντι anti-dumping. Ε, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε το θέμα αυτό και να συζητήσουμε ε, για την καλύτερη διαμόρφωση της οικονομικής μας συνεργασία με την Κίνα τα προσεχή χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο Μπέντ Λάγκ εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε θα συνδέσω την παρέμβασή μου με αυτά τα οποία είπε ο κ. Κασπάρη στο τέλος. Ε, ελπίζω να, ε, συμφωνεί... Ε, η τοποθέτηση σας διαφέρει με την τοποθέτηση της Γερμανίας, που είναι εντελώς διαφορετική. Κύριε Επίτροπε, αναφερθήκατε στις δυσκολίες επικύρωσης των διμερών συμφωνιών στο επίπεδο των χωρών μελών. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι οι συμφωνίες αυτές είναι μικτές, έχουν οριστεί μάλλον ως μικτές ε, συμφωνίες και κατά πάσα πιθανότητα θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και σε μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες. Ποια είναι η δική στρατηγική έναντι του Συμβουλίου και ε, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν οι αρμοδιότητες συνθήκες της Λισαβόνας και η εμπορική πολιτική να μην ε, να έγκυται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην υπονομεύεται από μικτές ε, συμφωνίες. Ε, τρίτον, είδα, ε, βρήκα τη θέση σας σε σχέση με την περίπτωση του, σχέση με τον όσα έγιναν στον Μπαγκλαντές και, και τα όσα υπόθηκαν στην Ολομέλεια, θεωρώ ότι είναι θετικά και τα στηρίζω. Θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο σε μελλοντικέ εμπορικέ συμφωνίε να μην υπάρξουν πιο έντονες αναδιατυπώσει όσον αφορά της, ε, τη χάραξη των σχετικών ε, πολιτικών βάσει του μοντέλου των βελγικών επενδύσεων ή την, ε, της συμφωνίας με την Αμερική. Και ο τρίτος τομέας στον οποίο δεν αναφερθήκατε είναι η αναθεώρηση της ε, νομοθεσίας Λιόζ γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι ε, γιατί εκτιμώ ότι τους προσεχείς μήνες πρόκειται να προχωρήσετε εδώ. Ε, δεν θέλετε να υπάρξουν καθυστερήσεις. Η κυρία Κόχμεριν για την Άλντε. Um, <clears throat> Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε και πάλι εδώ. Είμαστε ευγνώμονες που δεν ξεχάσατε το ραντεβού μας και κάτι που είχατε πει πριν από κάποιο καιρό σε επώδυνες ακροάσεις που περάσατε μαζί μας ότι θα είσαστε ανοιχτό σε συνεργασία και διαρκή διάλογο με το Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που πληρώσατε την υπόσχεσή σας και με τα χρόνια δεν ξεχάσατε την υπόσχεση αυτή. Θα ήθελα να θίξω δύο στοιχεία και είμαι βέβαιη ότι και η Κάθριν σε λίγο θα περάσει σε περισσότερες λεπτομέρειες που εγώ τώρα μπορεί να μην προλάβω. Πρώτον, είπατε ότι ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις με τον Καναδά για τη συμφωνία ΣΥΤΑ. Αυτά είναι πολύ καλά νέα. Αλλά το έχω ξανακούσει τα τελευταία δύο χρόνια επανειλημμένως. Πόσο τελικό στάδιο είναι αυτό το στάδιο της περάτωσης. Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια οριστική ημερομηνία για το πότε επιτέλους θα δούμε τη λήξη των διαπραγματεύσεων και να το γιορτάσουμε κιόλα. Και μάλιστα ποια ζητήματα παραμένουν εκκρεμή ακόμη. ποιε είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες και πού παραμένουν διαφωνίες στις συζητήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Κάτι άλλο. Και κάτι άλλο που το είπαν και ο κύριος Λάγκια και ο κύριος Κάσπαρη. Οι συζητήσεις μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα μέτρα κατά της Κίνας. Ακούσαμε έναν σωστό μάλλον υπολογισμό. 15 είναι τα κράτη-μέλη που δεν είναι ικανοποιημένα με το να ληφθούν μέτρα κατά της Κίνας, όπως τα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που στηρίζεται από 6 μέλη τουλάχιστον, ενώ κάποια απέχουν από την τοποθέτηση. Το Συμβούλιο πρόκειται να αποφασίσει. Ε, αναρωτιέμαι, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Τι θα γίνει αν έχουμε τέτοιου είδου ισορροπίε μεταξύ 100 και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια είναι η άποψή σα γι' αυτό και πείτε μα και μερικέ λεπτομέρειε για δύο ακόμα τομεί οι δασμολογικές διατάξεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πολύ γρήγορα αποφασίστηκαν και ε, επιβλήθηκαν προσωρινή δασμή. Γιατί έγινε αυτό και ποιες ε, ε, έσωθεν πληροφορίες έχετε για το, την εξέλιξη του όλου θέματος. Μπορείτε να μοιραστείτε κάτι μαζί μας από όσα ξέρετε. Διότι από τη μια η ανάλυση δεν έχει ολοκληρωθεί, από την άλλη ακόμα να λαμβάνονται συγκεκριμένα χειροπιαστά μέτρα. Και για τις τηλεπικοινωνίες. Νομίζω δεν βρισκόμαστε σε ένα κατάλληλο νομικό κλίμα εντό εισαγωγικών, διότι έχουμε μια καταρχήν απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαντάζομαι ότι η Επιτροπή του ΠΟΕ θα τοποθετηθεί σχετικά. Οπότε, αυτή καταρχήν απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν την έχει ενεργοποιήσει. Τι σημαίνει αυτό. βλέπετε να υπάρχει αντίφαση με το προηγούμενο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη να της ανατεθεί εντολή, διαπραγματευτική εντολή για επενδυτική συμφωνία με την Κίνα. Ταυτόχρονα τα, μέσα, τα μέτρα αυτά που ίσως δεν γίνονται αντίληπτα ως ε, μέτρα που διευκολύνουν το άνοιγμα του εμπορίου με τους Κινέζους εταίρους. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Θα ξανάρθουμε στην ομάδα σας στο δεύτερο γύρο. Ε, επόμενος, ο κύριος Κάμπελ, συντηρητική και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, από την τελευταία σας προσέλευση εδώ Ξέρω ότι έχετε κάνει μια εξαιρετική παρέμβαση στι βρετανικέ πολιτικέ. Από του Βρετανού βουλευτέ δεν ξέρουν τίποτα για την Ευρώπη και του προειδοποιείτε, παραθέτω, ότι θα γεννήσουν καταστροφέ που θα συμπαρασύρουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ θα χάσει τεράστια εμπορικά ωφέλη. σω με τίμημα δεκάδε χιλιάδε θέσει εργασία. Αυτό το είπατε στι 6 Μαου. Λέτε ότι χρειαζόμαστε αποφάσεις βασιζόμενοι σε γεγονότα και αριθμούς και όχι Πληροφορίε. Αλλά αφού κάνατε αυτή την παρέμβαση, για πείτε μου το εξή. Εάν η Βρετανία θεωρητικώ ε, οργάνωνε δημοψήφισμα το 2016-2017 και ψήφιζε να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μα λέτε ω Επιτροπό ε, Επιτεμπορίου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ανήμπορη πλέον να διαπραγματευτεί εμπορικέ συμφωνίε με του μεγαλύτερου πελάτε σα και μάλιστα το μεγαλύτερο από όλου που είναι η Βρετανία, 4 δι αγαθά και υπηρεσίες εισάγουμε από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση των 26, 26, 5 μάλλον δις ετησίω. Και επίσης, δεν θα διαπραγματευόσασταν καμία εμπορική συμφωνία με κάποια από χωρών μέλος. Γιατί δεν κάνετε με τις ΗΠΑ το ίδιο με την Συμφωνία Ελεύθερων Συλλαγών που έχετε κάνει με την Ελβετία, την Ορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί ε, είχατε, γιατί λοιπόν κάνατε αυτή την βία παρέμβαση στην Βρετανική πολιτική βασιζόμενη σε έναν τέτοιο μύθο. Ευχαριστούμε η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Έχω αρκετέ ερωτήσει, αλλά θα προσπαθήσω να τι συντομεύσω. Αναφέρατε την Κολομβία. Υπήρξε ο δικός χάρτη για το Περού, την Κολομβία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλε πτυχέ και διερωτώ με. Μπορείτε να μα πείτε πώ θα λειτουργήσει στην πράξη, Ποιο θα υπεύθυνο για την υλοποίηση αυτού του δικού χάρτη, όλων των δικών χάρτεων. Πότε να περιμένουμε την πρώτη καταγραφή των αποτελεσμάτων μετά την υλοποίηση του εμ, χάρτη. Αναφέρεται και το Μιανμάρ και την υποβολή εκθέσεων. Θα υπάρξει έκθεση προόδου για τα εργασιακά δικαιώματα και πρότυπα κτλ. πριν περάσουμε στην επόμενη φάση του καθεστώτος προτιμησιακού ε, το 2014 για το GTI να πω ότι είναι σημαντικό το Ευρωκοινοβούλιο είναι σημαντικό να λάβει πλήρως το ρόλο του ως ε, νομοθέτης και να μην μείνει στο περιθώριο όπως σε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, γιατί εδώ τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Θέλουμε να έχουμε έναν πλήρω και ενεργό ρόλο εδώ. Επίσης, να πω ότι εδώ πραγματικά στηρίζω το ΕΛΚ για το θέμα της Κίνας. Δεν θα πρέπει να παραδοθούμε, ούτε να υποχωρήσουμε ως προς τις Ηνωμένε Πολιτείες αναφέρατε ότι η διαφάνεια είναι άκρο σημαντική. Ακόμα και σε ιδιαίτερες συνθήκες. Πιστεύουμε παρόλα αυτά ότι η εμπορική συμφωνία με τι Πολιτείε είναι σημαντική ώστε να υπάρξει εφόσον μάλλον υπάρξει διαφάνεια στι ενεξελίξεις διαπραγματεύσει, κάτι που έπρεπε να συμβαίνει και προηγουμένω. Εάν δεν υπάρχει, δεν θα πετύχουν οι διαπραγματεύσει. Τι θα κάνετε λοιπόν με τη διαφάνεια, πώ θα ενημερώνετε του πολίτε αλλά και του βουλευτέ για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και την εντολή σα. Και επίση, σημαντικό είναι να λάβετε σοβαρά τι ανησυχίε μα για τα οπτικοακουστικά λόγω χάρη, αλλά και για τα υπόλοιπα πρότυπα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που δεν θέλουμε να διακυβευτούν εξαιτία τη συμφωνία με τι ΗΠΑ. Εδώ χρειάζεται η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου προκειμένου αυτά να ακουστούν. Είμαι βέβαιη ότι εδώ υπάρχει ουσία. Ε, για τον Μπαγκλαντέ, το Κοινοβούλιο ψήφισε πριν από δύο συνόδου ολομέλεια να προβλεφθεί να προβλεφθούν κανόνες κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και εκεί, δεσμευτικοί κανόνες. Τι σκοπού έχετε για να εφαρμοστεί αυτό, μια και αναφέρετε το υποχρεωτικό στάδιο. Και επειδή αναφέρετε και το είπα, έχετε δει την έκθεση Επιτροπής ε, ΙΝΤΑ Αποστολή μάλλον και αντιπροσωπείας ΙΝΤΑ οι οποίοι μελέτησαν το θέμα αυτό και είδαν ε, ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Και στην Ινδία, ποια είναι η κατάσταση εκεί πέρα. Θα ήθελα λίγα λόγια και γι' αυτό. Πρόεδρος, δεν βλέπω κανέναν από, τον Γκουε, από την ΚΟΕ, τελευταίο στο γύρο αυτό, για την Ευρώπη της Δημοκρατίας και Ελευθερίας, ο κ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους και τον Επίτροπο που ήρθαν σε αυτή τη συνάντηση. Ε, εκφράστηκε με τη συνήθι αφήνεια και διαβιά του. Ήθελα εδώ να θέσω δύο ερωτήσει για θέματα που δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Πρώτα απ' όλα, για τα σχόλιά σας για το Ηνωμένο Βασίλειο το σημερινό τοπίο και εφόσον από τότε μάλλον που το Ηνωμένο Βασίλειο προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1973 έχουμε ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα 573 εκατομμύρια διστερλίνες αυτό είναι ένας αριθμός που ανέφερα και σε μια ομιλία μου το Σεπτέμβριο έχουμε φτάσει πλέον στο Μάιο και είναι σίγουρο ότι έκτοτε το έλλειμμα θα έχει αυξηθεί αυτό που είπατε λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τι ήταν προσωπική πρόβλεψη από πλευρά σα. Ή μιλήσατε επισήμω ω ε, επίτροπο ή εκ μέρου τη Επιτροπή συνολικά του Κολέγιου των Επιτρόπων. Βάσει των όσων είπατε, ήταν δική σα πρόβλεψη. Μια και μιλάμε υποθετικά ούτω ή άλλω πάντοτε για το μέλλον. Ήταν δική σα πρόβλεψη ότι αν το Ηνωμένο Βασίλειο φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει την ίδια ή παρόμοια εμπορική συμφωνία ελευθερών συναλλαγών όπως αυτή που υπεγράφει με το Μεξικό, την Νότια Κορέα και την Κολομβία ή τέλο πάντων που προγραμματίζεται με την Κολομβία και τους υπόλοιπους. Δεύτερη ερώτηση τώρα. Για τους δασμούς που έχουν να κάνουν με, τα φωτοβολταϊκά, με τους φωτοβολταϊκούς πίνακες που κατασκευάζονται στην Κίνα σε τέτοιες ε, δυσχερείς οικονομικές συνθήκες. Βλέπω ότι οι Γερμανοί βουλευτές δεν αντιδρούν ή δεν έχουν αντιρρήσεις που είναι διαφορετικό θέμα. Είναι τα 14 τα κατημέλη που έχουν αντιρρήσει εδώ και σε τέτοιες οικονομικές συνθήκες 17 κράτη-μέλη εμποδίζουν την πρωτοβουλία αυτή. Να ρωτήσω λοιπόν, εάν πάνω από τα μισά κράτη-μέλη διαφωνούν πλειοψηφία και αριθμητική αλλά και ως προς τον πληθυσμό τους. Αυτό δεν σας δίνει την, το ηθικό κύρος και την εξουσία να ξεκινήσετε μια εκστρατεία τιμωρητικών ε, δασμών 47% κατά της Κίνας και επιβεβαιώνεται ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι ίδια πρωτοβουλία. Έχει δηλαδή αναλυθεί χωρίς καμία προηγούμενη έγκριση από τα κρατη Δεν είναι αυτό που ένας Βρετανός δικηγόρος θα έλεγε στο δικαστήριο κάτι τελείως αυθαίρετο που δεν έχει καμία στήριξη από τα κρατη Κάθε νόμος, μάλλον κάθε δράση οδηγεί και σε αντίδραση. Αυτό είναι νόμος της φυσικής αλλά είναι και της πολιτικής και ισχύει για τους εμπορικούς δασμούς. Παράδειγμα, οι εταιρείε στην εκλογική μου περιφέρεια, γιατί έχουμε σημαντικέ βιομηχανίε, που εγκαθιστούν, τοποθετούν πίνακε, θα πληγούν από την εφαρμογή αυτών των δασμών. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για θέσει εργασία στην κατασκευή. Εάν θε, ε, σώστε θέσει εργασία ε, στον κατασκευαστικό τομέα, θα εμποδίσετε στην τοποθέτηση και τη διανομή να δημιουργηθούν περισσότερε ή να καταστραφούν κάποιε εκεί. Αυτό είχα να παρατηρήσω και σα ευχαριστώ για τον χρόνο σα και την προσοχή σα. Πρόεδρο. Δεύτερο ε, γύρο για τα επόμενα αιτήματα. Uh, ο Επίτροπος πρέπει να απαντήσει σε αυτά και μετά να ακολουθήσει ο δεύτερο γύρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορεί να υπάρξουν και πρόσθετα ερωτήματα, αλλά μπορεί κάποια από αυτά να έχουν απαντηθεί όταν θα έχω ολοκληρώσει την ε, πρώτη μου απάντηση. Έχω δε την εντύπωση ότι ήδη ε, ρωτήσατε σχεδόν τα πάντα. Τέλο πάντων, σε ένα κοινοβούλιο βέβαια δεν μπορεί κανεί να γνωρίζει. Μην υποτιμάτε τη δυνατότητα τη Επιτροπή και την ικανότητα των μελών να κάνει ερωτήσει, λέει ο Πρόεδρο. Για τι ΗΠΑ, ελπίζω να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τον ήλιο τη διαπραγματεύση. Νομίζω ότι υπάρχουν εύλογε πιθανότητε να συμφωνήσουμε μέχρι τι 14 Ιουνίου για την εντολή των διαπραγματεύσεων στο Λουξεμβούργο. Δεν θα επεκταθώ ε, σε συζήτηση για τα οπτικοακουστικά. Αν δείτε όμως τις τρεις κόκκινες γραμμές που ανέφερα και στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα μπορούσε να συμβεί στις διαπραγματεύσεις που θα αντέβαινε στην πολιτισμική πολυμορφία. Πραγματικά δεν το βλέπω, σας μιλώ ειλικρινά και βέβαια ότι έχει να κάνει με την πολιτιστική και πολιτισμική πολυμορφία θα πρέπει να γίνει δεκτό ομόφωνα. Ειλικρινά λοιπόν έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Τώρα το, τα πόσο θα καταλήξουμε σε λύση αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά τουλάχιστον μπορέσουμε να τα συζητήσουμε. Υπάρχει μια πολύ γρήγορη εξέλιξη στον τομέα αυτό. Έρχονται κατακύματα κύματα εξέλιξη, δύο στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Από την Apple, από την ε, ε, Google, το Netflix ε, και όλα τα άλλα πρώτα που φτάνουν στο καταναλωτή. Άρα όλα αυτά εντάσσονται σε ένα πολύ πιο ευρύ πρόβλημα. Το θέμα είναι πώ θα μπορέσουμε να ελέγξουμε ε, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κάποιο άλλο ενδεχομένω να ελέγξει, να παρακολουθήσει τι εξελίξει αυτέ και στο μέλλον. Α έχουμε τουλάχιστον δυνατότητα να τα συζητήσουμε με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Θα δούμε όμως ε, στην εντολή τι θα συμπεριληφθεί. Πάντως κατενόησα το μήνυμα του Κοινοβουλίου. Ούτε εσείς ούτε τα μέλη σας, κύριε Πρόεδρε, της Επιτροπής είναι υπεύθυνοι. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση στην Ολομελία. Όχι μόνο μέλη της δικής σας Επιτροπής. Ε, είναι κρίμα, γιατί από το 80 στο 94 αυτό βλέπουμε. Στην Ολομέλεια μιλούν οι ίδιοι οι οποίοι μιλούν και στην ε, Επιτροπή. Και πλένε τα προβλέψιμα ουσιαστικά. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει ευρύτερη συμμετοχή και από άλλους βουλευτές. Έτσι είναι η ζωή όμως. Κίνα. Στο Σώμα των Επιτρόπων έχω προτείνει μια εντολή, ένα σχέδιο εντολής. Το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει από αυτή τη εντολή. Το σχέδιο εντολής αφορά την προστασία των επενδύσεων και την πρόσβαση στην αγορά. Πάντοτε ε, καθιστούμε σαφές στην Κίνα ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές, αλλά θα πρέπει σε αυτές να περιλαμβάνεται και το σκέλος της πρόσβασης στις αγορές. Δύο φορές συγκεκριμένα τα συμπεράσματα των διασκέψεων κορυφής με την Κίνα ανέφεραν ότι εν λόγω διαπραγματεύσεις θα πρέπει να αφορούν θέματα ενδιαφέροντος και για τις δύο πλευρές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το και προς τις δύο πλευρές δηλαδή μπορεί ε, θέματα για τα οποία δεν συμφωνεί κατά ανάγκη και η άλλη πλευρά να μπουν στην, ε, στις διαπραγματεύσεις. Αυτό το οποίο θα ήθελα να δω από την Κίνα και να ξέρω είναι αν και αυτοί θα σημειώσουν πρόοδο ε, με ό,τι αφορά τη δική τους εντολή λένε ότι είναι έτοιμοι, ότι κάνουν πρόοδο. Πού βρίσκονται όμως ακριβώς, δεν ξέρουμε. Έθεσα λοιπόν το θέμα στο Συμβούλιο. Αλλά όταν καταλήξουμε νομίζω σε σχέση με την εντολή, δεν νομίζω ότι θα είναι τελικά τόσο δύσκολα τα πράγματα με το Συμβούλιο και τότε θα έχουμε και μια πιο σαφή εικόνα για το τι έχουν στο μυαλό τους και οι Κινέζοι. Κάτι που οφείλω να πω ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να μάθουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, διμερείς ε, συνθήκες ε, επενδύσεων, δεν θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία σύναψης μια συμφωνίας επενδύσεων, προστασίας επενδύσεων με την Κίνα. Επισήμως έγινε η σχετική πρόταση στη διάσκεψη κορυφής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους δύο Προέδρους, Φανδρομπέ και Μπαρόζο. Επομένως αυτή τη χρονική στιγμή δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να έχουμε διαπραγματεύσεις για μια διμερή συνθήκη επενδύσεων ενός κράτους σημαίνει δηλαδή της Ένωσης με την Κίνα. Ούτε νόημα θα είχε και μπορούμε, έχουμε την εξουσία να αντιταχθούμε και αυτό θα πράξουμε. Um, <coughs> was the problem with You still remember? You, you δεν θυμάμαι τι με ρωτήσατε. Ο κύριος Κάσπαρ. Όχι, δεν αφορούσε η ερώτησή μου ε, μέλη της Ένωσης και την Κίνα, αλλά το Βιετνάμ, το Καζακστάν και ένα μέλος της Ένωσης. Απάντηση, δεν έχουμε λάβει αιτήματα τέτοια μέχρι τώρα. Με το Βιετνάμ είναι μέρος των διαπραγματεύσεων για μια επενδυτική συνθήκη. Είναι θέμα πλέον να επαναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στα κρατημέλη μεμονωμένα σε ό,τι αφορά την ε, ανακατανομή των ε, ανθρώπινων πόρων. Αυτό το μείον 1% δεν μας αφορά. Άρα η γάμα δέλτα η δικιά μας έχει μια καλύτερη μεταχείριση από άλλες προς το παρόν. Δεν είχαμε βέβαια μέχρι στιγμής πολύ φορτωμένη μέσα διάταξη. Αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε και λίγο παραπάνω προσωπικό. Κάποιος σίγουρα πρέπει να χάσει κάποιες θέσεις εργασίας. Και ορισμένοι νομίζουν ότι τον έχουμε στον τόπο στις θέσεις εργασίας είναι και ένα ε, κληροδότημα που αφήνουμε. Τέλος πάντων. As much as we can. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε ό,τι καλύτερο. Για τους ε, ολιακούς συλλέκτες υπάρχουν ε, πολλά θέματα στην Επιτροπή κατά του dumping Νομίζω είναι 14-15 κρατημέλη αυτά τα οποία έχουν καταψηφίσει, από ό,τι ξέρω. Βέβαια, γνωμοδοτούν ουσιαστικά, δεν αποφασίζουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει αν θα επιβάλλει ή όχι κάτι. Δεύτερον, όταν βλέπετε την σύνθεση, δηλαδή και δείτε ποιοι ψήφισαν υπέρ, ποιοι ψήφισαν κατά και ποιοι απήχαν, Εύχομαι εδώ και στους ε, συναδέλφους ε, σας πέρασαν τις ερωτήσεις. Δεν έχουμε τη σχέση 15 προς 12. Ξέρετε ότι υπάρχει και στάθμιση ψήφων. Δεν λέω δεν το γνωρίζετε, αλλά εκινάται από ασφαλμένο συμπέρασμα, εσφαλμένη υπόθεση. Γιατί πρέπει να δούμε ποια κράτη-μέλη είναι μεγάλα ή μικρά και τι στάθμιση ψήφων υπάρχει. Η Κομισιόν έχει να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις ε, διαδικασίες. Και πάντοτε το έλεγα πολύ ξεκάθαρα. Το είπα και στον Κινέζο Υφυπουργό, δημοσία το είπα και χθε σε Ιάπωνες δημοσιογράφους. αν ασκούν πίεση σε κάποιο μεμονωμένο κράτος, δεν πρόκειται να με εντυπωσιάσουν, δεν μου καίγεται καρφί. Το αν είναι ένα ε, μικρό νησιωτικό κράτος ή αν είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, εμένα δεν με αφορά καθόλου, ας ασκήσουν, αγίως προσπαθήσουν να ασκήσουν πιέσεις, θα χάσουν το χρόνο τους μαζί μου. Ας το προσπαθήσουν. Και αν δείτε τη διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας είπα, ότι απλά περί γνώμης πρόκειται. Αν εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Γιατί σας διαβεβαιώ ότι κάτι δίαν αυτοί που ακριβώς καταψηφίζουν δεν λένε ακριβώς τα ίδια. Και κάποια κράτη φοβούνται να ψηφίσουν όπως πιστεύουν ότι θα έπρεπε να ψηφίσουν. Και αυτό δεν είναι καλό. Εγώ δεν θα τα δεχθώ αυτά. Ούτε θα υποχωρήσω. Μπεντ Λάγκε. Δεν θα σχολιάσω για την Κίνα, τη θέση για την Κίνα. θα μπορούσα να πω κάτι παραπάνω, αλλά δεν θα το κάνω. γιατί οι πολιτικές απόψεις δεν είναι πάντοτε απλές. Για τον Παγκλαντές. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Αλλά αυτό να γίνει και στον Παγκλαντές και στη ΣΥΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ και εγώ είμαι πρόθυμος, αλλά και οι ιδιωτικέ εταιρείε. Θα πρέπει και αυτές να συμμετάσχουν. Και φυσικά θα συνεργαστούμε και πρέπει να συνεργαστούμε τις αρχές του Μπαγκλαντές, κάτι που δεν είναι εύκολο, γιατί έχουμε να κάνουμε με χιλιάδες επιχειρήσεις σε αυτήν την αψόμενη χώρα. Έχουμε μια διαδικασία, το θέμα είναι να πάρει τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είμαι διατεθειμένος να δεχτώ ότι θα έχουμε εμπόριο μαζί τους μόνο αν παίρνουν 30 40 δολάρια το μήνα. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μια σαφή κατεύθυνση και να δούμε τι κάνει τον Μπαγκλαντές για τους φτωχούς αυτούς ανθρώπους. Κοινή είναι η ευθύνη και η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και εμείς έχουμε ευθύνη. Και θα προσπαθήσουν να σημειώσουν μια ουσιαστική πρόοδο. Έγινε μια ερώτηση από την κυρία Κέλλερ για το Μπαγκλαντές, μια καλή ερώτηση. Ε, οτιδήποτε εκτός από όπλα. Και αν δούμε τους όρους που διατυπώνονται σε αυτή τη συμφωνία Everything But Arms, δεν είναι τόσο... δεν υπάρχει τέτοιο εύρος. Και το σκεπτικό είναι ότι όταν επιβάλλονται υπερβολικοί όροι, τότε οι, λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες δεν μπορούν να συνεργαστούν μαζί σας. Θα πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια ισορροπία. Για παράδειγμα, εγώ το εξέτασα και ο αριθμός των συμβάσεων ε, με την ILO ε, δεν είναι εξαντλητικό. Όταν θέλουμε να ληφθεί δράση, δράση, γιατί καταρχήν θα πρέπει να τους δώσουμε κάποια ευκαιρία να επιδείξουν κάποιες βαλίστες πρακτικές. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε μόνο στη βάση μιας έκθεσης του ILO. Και η παρούσα έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας λαμβάνει υπόψη της ε, μια διαδικασία εμείς συνήθως ε, βασιζόμαστε στα ευρήματα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και όταν αυτοί καταλήξουν στο αποτέλεσμα ότι υπάρξει σοβαρή παραβίαση αρκετών προϋποθέσεων, ε, θα ήθελα να διασφαινίσω ότι είμαι κατά των περιορισμών στις εισαγωγές. Εγώ αναφερόμουν ε, στους δεσμευτικούς κανόνες για το CSR, για την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Εκεί αναφέρθηκα. Ναι, αλλά έχουμε τις δύο πλευρές. Εσείς αναφέρεστε στην κοινωνική εταιρική ευθύνη και εγώ πιστεύω ότι πράγματι οι επιχειρήσεις ε, φέρουν μια ευθύνη. Ε, και ε, θα πρέπει να είναι δεσμευτική αυτή η όρη. Νομίζω ότι πραγματικά έχουν, φέρουν μια ευθύνη για την αλυσίδα εφοδιασμού και κατά πάσα πιθανότητα βεβαίω δεν είναι δυνατόν να γίνουν έλεγχοι σε όλου του υπεργολάβου κλπ. Αλλά δεν είναι μικρομεσαίε επιχειρήσει, είναι ε, μεγάλε εταιρείε και θα πρέπει να κάνουν τι κατάλληλε επενδύσει ούτω ώστε να είναι σωστή η αλυσίδα εφοδιασμού και να ελέγχεται, να υποβάλλεται σε συνεχεί ελέγχους. Εγώ πάντοτε υπήρξα ιδιαίτερο ε, αυστηρό σε αυτό. Ε, και επίση και για τα μέταλλα τα οποία προέρχονται από ζώνες ένοπλης σύραξης. Όσον αφορά τη δυτή χρήση, θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το διέξοδο ε, μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου μέσω του Omnibus και αν ε, δεν γίνει αυτό δεν μπορούμε να προτείνουμε μια μεταρρύθμιση του συστήματος ε, διτής ε, χρήσης ούτως ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα τηρώντας τις προδιαγραφές ασφαλείας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια συμφωνία, μια ολοκλήρωση του Omnibus και στη συνέχεια θα υποβληθεί σχετική πρόταση. Κυρία Κοχμερίν, ε, θέσατε το ερώτημα για τον Καναδά. Είπατε ότι ελπίσαμε για κάποιο καιρό ότι θα ολοκληρωθεί μια τέτοια συμφωνία. Και εγώ ίδιος είχα αυτή την ελπίδα και όταν πήγα στην Οτάβα που έκανε πολύ κρύο παρεπιπτόντας, όχι στην αίθουσα συνεδριάσεων αλλά έξω Χωρίς να θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, εξελίσσεται μια συζήτηση. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες, αλλά βεβαίως λεπτομέρειες μπορούν να είναι πολύ καθοριστικές στη σύναψη μιας συμφωνίας και γίνεται μια συζήτηση για την αναλογία μεταξύ φρέσκου και κατεψυγμένου κρέατος όταν εξάγεται κρέας στην Ευρώπη μπορεί να είναι φρέσκο ή κατεψυγμένο και αυτό έχει μεγάλη διαφορά στην τιμή και υπάρχει λοιπόν μια σχετική συζήτηση. Αυτή δεν είναι ε, πολιτική υψηλού επέδου αλλά ωστόσο είναι σημαντική αυτή η διαφορά και έχω λοιπον μια σχετικη συζητηση αυτη δεν ειναι ένας ειδικό για το θέμα αυτό, όχι δεν ήξερα ότι υπάρχει μια διαφορά. Επίσης, ε, γίνεται μια σύντηση για ορισμένε διαστάσει των δημοσίων ε, συμβάσεων. Ε, κατά τα λοιπά, νομίζω έχουμε συμφωνήσει. Θα δω τον Υπουργό του Καναδά μεθαύριο στο Παρίσι, γιατί υπάρχει μια διευπουργική συνάντηση εντός του ΩΣΑ και νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε μια συμφωνία. Αλλά για τις τηλεπικοινωνίες αυτό το οποίο κάνουμε είναι να λάβουμε την απόφαση ε, ότι είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε, να συνεχίσουμε εδώ. Και η διαδικασία για τα φωτοβαλταϊκά ε, βασίζεται σε κάποιες ε, προσφυγές εκ μέρους κυρίως γερμανικών εταιριών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η νομική διαδικασία για την Telecom θα είναι ε, μια διαδικασία και υπήρξε μια ομόφωνη απόφαση σχετικά με αυτό και θεωρώ ότι αυτό έχει επίση μια σημασία. Λήφθη εδώ ομόφωνα μια απόφαση και όχι ως αποτέλεσμα άσκησης ε, πίεσης. Ε, και σήμερα δίνουμε στους Κινέζους αρκετό χρόνο ούτως ώστε να διαπραγματευτούν μια λύση αλλά ανεπόκειται σε αυτούς και αν όχι θα ενεργοποιήσουμε αυτή τη ε, διαδικασία, ποινική διαδικασία. Ε, και αυτή είναι μια σημαντική ε, συζήτηση με την Κίνα. Νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική συζήτηση περιμπορίου αυτή τη στιγμή εκτός από αυτή που γίνεται, επεκτελείστε με τις ΗΠΑ αλλά σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Δεν πρόκειται ε, για μία διαμάχη. Εδώ. Αλλά αυτή είναι μια, ένα θέμα χρήσιμη σημασία. Γιατί όταν αρχίσει να ανταγωνίζεται εμά η Κίνα, είτε το επιθυμούν είτε όχι, θα πρέπει να σέβονται ένα πεδίο ισότιμων όρων ε, και για την κινητή τηλεφωνία και για τις, τα φωτοβολταϊκά κλπ όλες ε, ε, αυτές οι εταιρείε ε, είναι κρίσιμη σημασία. Έχουν το δικαίωμα να μας ανταγωνίζονται, αλλά θα πρέπει να το κάνουν τηρώντας συγκεκριμένους κανόνες. Κύριε Κάμπελ, Μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά εμένα μου αρέσουν οι Βρετανοί πολιτικοί, έχουν πολύ στυλ. Και εσείς ειδικά, εάν φεύγατε θα μας λείψετε. Αλήθεια, αλήθεια. Δεν σας κοροϊδεύω. Θα μας ε, λείπατε γιατί δίνετε ένα ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη τρόπη στις συζητήσεις. Είστε τόσο θυμωμένος ή μάλλον φαίνεστε θυμωμένος χωρίς να είστε και μάλιστα με χιούμορ. Μ' αρέσει εμένα. understand anything about Δεν είπα ότι οι Βρετανοί δεν έχουν καταλάβει τίποτα για την Ευρώπη. Καθόλου δεν είπα κάτι τέτοιο. Μπορώ να πω την άποψή μου για τη Βρετανική πολιτική, γιατί και εσείς μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είστε. Δεν σημαίνει ότι είναι άποψη του σώματος των Επιτροπών. Δεν εξέφρασα συνολικά τη δική τους την ε, άποψη αλλά κατεδία νομίζω περισσότεροι συνάδελφοί μου θα συμφωνούσαν μαζί μου. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Τώρα το αν τα λέω ω επίτροπος ή ω άνθρωπος, ελπίζω να πιστεύετε στην ελευθερία του λόγου. Τι θα ήταν το κοινοβούλιο χωρίς ελευθερία του λόγου. Τέλος πάντων. Ε, πώς έγινε όλο αυτό. Έφτασα στο Παρίσι και στο διπλανό τραπέζι. Ήταν ένας συντηρητικός βουλευτής του κοινοβουλίου και αρχίσαμε να τα λέμε. Και ήταν ευρωσκεπτικιστής και προσπάθησα να τον πείσω, να τον πάρω με το μέρος μου. Σχεδόν τα κατάφερε. Όταν μέχρι να φτάσουμε στο γλυκό. Διότι αλήθεια είναι ότι, ότι υπάρχουν πολλές παρανοήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά προσπαθούσα να εξηγήσω και ως πολιτικός δεν είμαι κανένας ψηλόβαθμος δημοσίου υπάλληλο, πολιτικός είμαι. Ε, είπατε, είναι άποψή μου. Δεν θα με υποχρεώσετε να σας πω και συγγνώμη όμως. Τώρα το αν θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, δεν είναι θέμα αυτό τώρα. Δεν είναι αυτό το θέμα μάλλον. Είστε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ώρα. Ελπίζω και απέφχομαι την αποχώρησή σας. Οπότε το να συζητάμε υποθετικά θέματα ενώ υπάρχουν τόσα πραγματικά ζητήματα που θα πρέπει να σας απασχολούν και στα πρέπει να απαντήσω, έμαθα για μια καινούργια λέξη, το φρόλικ. Μου το εξήγησε η βοηθός μου. Χορός είναι, έτσι. She says it's une danse frivole. Very nice. So frolic. Um... Είναι ένας ε, χαρούμενος ε, χορός. Τέλος πάντων, ο Ρόδο Ντάρτμουντ μίλησε για μεγαλύτερο κύρος. Αυτά μου αρέσουν ακόμη πιο πολύ από αυτά που ο κύριο Κάμπελ. Δεν με ενόχλησε καθόλου. Κυρία Κέλλερ, για τον οδικό χάρτη. Ακριβώς αυτό συμφωνήσαμε, σωστά τα λέτε. Θα δούμε πότε θα φτάσει η πρώτη έκθεση, αλλά μάλλον πριν από το τέλος αυτής της θητείας. Συμφωνώ μαζί σας το ίδιο και για το Μιανμάρ. Πρώτη έκθεση πριν από το τέλος της θητείας, λογικά. Για το TDI, Μα εδώ μπορεί να αναλάβει πλήρω το ρόλο του Ευρωκοινοβούλιο και μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για το τι θα περιλαμβάνει. Ίσως είναι κάπως πιο δύσκολες οι διπλωματεύσεις με το Συμβούλιο, αλλά δεν νομίζω με το Κοινοβούλιο Λέτε να μην ε, υποχωρήσω με την Κίνα, για την Κίνα μάλλον, εν, μπροστά στους Κινέζους. Δεν πρόκειται να το κάνω. Για το Τρινιτάτ και τον Πάγκο. Δεν την ξέρω την έκθεση, δεν την έχω δει. Θα το δούμε όμως. Δεν την ξέρω και απ' έξω. Και για τη διαφάνεια, ευχαριστώ να πάμε όσο μακριά θέλετε σε αυτό το τομέα. Νομίζω οι συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες κανονικά θα έπρεπε να μας επιτρέπουν να είμαστε διαφανέστεροι από τις άλλες διαπραγματεύσεις. Αρκεί βέβαια να συμφωνήσουν από την πλευρά τους και οι Αμερικανοί, αλλά εγώ θα τους το ζητήσω. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ διαφάνεια. Τα επιχειρήματα είναι σοβαρά. Μπορεί να χρειαστεί στο τέλο να καταλήξουμε σε συμφωνία μέσω διαιτησία. Κάποια διαμεσολάβηση τέλο πάντων μπορεί να χρειαστεί για να βρεθεί σωστή ισορροπία. Αλλά θα είναι πολύ ανοιχτότερη συζήτηση και ανοιχτότερε διαπραγματεύσει από ότι με άλλε χώρε, όποια και αν παράδειγμα. Οι δυσκερέστερε διαπραγματεύσει που είχαμε θα ήταν με μια χώρα που δεν είναι πολύ δημοκρατικό κράτος, λόγω χάρη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τη διαφάνεια. Νομίζω το έχω καταστήσει σαφές. Ποια είναι η άποψή μου για πολλά ζητήματα. Βεβαίω, δεν διαπραγματεύομαι μόνο μου, υπάρχουν και οι απέναντι. Οι συνομιλητέ. Αυτή τη στιγμή οι συνομιλητέ μου επιβεβαίωσαν. Πρέπει μάλλον να επιβεβαιώσουν προηγουμένω. Αλλά ε, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Κανένα. Και υπάρχει και διαφορά μεταξύ του να είναι κανείς διαφανής και να λέει ε, και να αποκαλύπτει ποια χαρτά του μένουν στο μανίκι. Ε, δεν το κάνει καν αυτό ένας καλός διαπραγματευτής, θα κρατάει. Στο μανίκι του. Λογικό είναι. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πρόεδρος, συνάδελφοι, τέλειωσε ο χρόνος. Time out. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιοι δεν πρόλαβαν να θέσουν τις ερωτήσεις τους, αλλά την επόμενη φορά θα είναι πρώτες στο κατάλογο. Σας ευχαριστώ και πάλι, Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πολύ. Yes, definitely. from Chinese. Full support.